we better, we better get... Αγαπητοί συνάδελφοι, ας ξεκινήσουμε και πάλι. Έχουμε ακόμα αρκετό δρόμο. Πρώτα απ' όλα, καλωσορίζουμε εδώ την κυρία Λίβια Γιαρόκα, τη συνάδελφό μας, που θα μας ενημερώσει για το θέμα το Ρώμα για πρώτη φορά. Ξέρετε ότι έχουμε συμπεριλάβει αυτό το θέμα στην ημερήσια διάταξη σήμερα, ώστε να ακούσουμε και από μια ομάδα από το London School of Economics, που τους τελευταίους μήνες δούλεψε πάνω σε μια μελέτη για μέτρα προώθησης του θέματος των ε, Ρώμα, πολιτών της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης, μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ακούσουμε σήμερα την προσωρινή έκθεση, γιατί η τελική θα έχει συμπληρωθεί δηλαδή μέχρι τις 15 Νοεμβρίου. Οπότε η ομάδα των μελετητών θέλει να ακούσει τα δικά σας σχόλια και τις δικές σας προτάσεις σήμερα. Μετά από την παρουσίαση αυτή του London School of Economics, θα ακούσουμε την εισηγήτριά μας, την κυρία Λίβια Γιαρόκα. Έχει ένα έγγραφο εργασίας που έχουμε ήδη κοιτάξει μια φορά. Τέλος. Όσον αφορά τη διαδικασία, περιμένουμε η διάσκεψη των Πρόεδρων να μας επιτρέψει να εκπονήσουμε έκθεση μάλλον θα εκπονήσουμε, να υποβάλουμε στην Ολομέλεια την έκθεση πρωτοβουλία μας. Χρειαζόμαστε αυτή την έγκριση, την οποία κανονικά η διάσκεψη των Προέδρων θα την δώσει στην επόμενη συνεδρίασή της. Συνεπώς, ακούμε την πρώτη παρουσίαση της μελέτης του London School of Economics. Καλώς ήρθατε. Ποιος από εσά θα πάρει το λόγο. Εσείς. Παρακαλώ. Έχουμε δύο μιλητές. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ. Είναι μεγάλη μου χαρά που βρίσκομαι σήμερα εδώ για να σας παρουσιάσω την προσωρινή μας έκθεση όσον αφορά μέτρα για την πρόθεση της κατάστασης των Ρώμα Ευρωπαίων πολιτών μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ονομάζομαι Βιλ είμαι επικεφαλής τμήματος στο London School of Economics. Και έχω μαζί μου και τη Ρομπέρτα Μπενίνη που είναι από την οργάνωση νομίσμα στην Πολωνία και τον Γορτ Τζόρνταν, ο οποίος είναι επίσης από το Πανεπιστήμιο. Αυτός ο τρίτος συνεργάτης δεν είναι εδώ μαζί μας σήμερα. Στην ομάδα μας έχουμε και τον Γιάννη Κάμπριελ που είναι εδώ από τις Βρυξέλλες και έχουμε και 12 εμπειρογνώμονες από τις χώρες ε, στις οποίες έγινε μελέτη και που καλύπτονται από τη μελέτη. Θα σας παρουσιάσω λοιπόν την μελέτη μας σε δύο τμήματα. Εγώ θα κάνω την πρώτη παρουσίαση, 10 λεπτά περίπου. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος για να μας δοθεί ευκαιρία να έχουμε και συζήτηση. Η Ρομπέρτα Μπενίνη στη συνέχεια θα σας παρουσιάσει τα συμπεράσματα και τις συστάσεις. Ευθύ εξ αρχή, επαναλαμβάνω, πρόκειται για την προσωρινή έκθεση, γιατί εξακολουθούμε τη δουλειά μα. Και γι' αυτό και θέλουμε πάρα πολύ να ακούσουμε τα δικά σα σχόλια. Θα μα βοηθήσουν πάρα πολύ να ολοκληρώσουμε αυτή τη μελέτη. Συμπεριλαμβάνονται 12 χώρες στη μελέτη. Έξι από αυτέ είναι από τι παλιέ χώρε. Η Γαλλία, η Γερμανία, η Ελλάδα, η Ιταλία, η Ισπανία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Οι άλλε έξι είναι νέε χώρε μέλη. Η Βουλγαρία, η Τσεχία, η Ουγγαρία, η Πολωνία, η Ρουμανία, η Σλοβακία. Έχουμε εκθέσει για την κάθε χώρα που παρουσιάζονται χωριστά. Καταλαβαίνω ότι δεν τις έχετε ακόμα. Θα τις έχετε όμως μέσα στις επόμενες ημέρες δείχνουν και αυτές οι εκθέσεις ότι είμαστε σε ένα προκαταρτικό στάδιο. Σας είπα ότι δεν πρόκειται για την τελική έκθεση. Λοιπόν, η παρουσίαση αυτή αποτελείται από τέσσερα τμήματα. Πρώτον, εισαγωγή που μιλάει για τις διάφορες έννοιες και για το πλαίσιο που ισχύει στην πολιτική. Το δεύτερο είναι μια πολιτική ανάλυση που αναφέρεται στον τομέα της απασχόλησης και της εκπαίδευσης. Γιατί, γιατί αυτά είναι πολύ βασικά θέματα όσον αφορά την ένταξη των Ρώμα και την βελτίωση της ε, ζωής τους. Στην πλήρη έκθεση περιλαμβάνουμε και την υγεία. Είναι και αυτός ένας τομέας πολιτικής που μας απασχολεί. Βέβαια είναι αλληλένδετες οι πολιτικές και των τριών αυτών τομέων. Οπότε μόνο αν έχουμε συνολική αντιμετώπιση, ολοκληρωμένη πολιτική και για τους τρεις αυτούς τομείς, μπορούμε να είμαστε σίγουροι για την επιτυχία. Το τρίτο τμήμα αναλύει τα νομικά μέσα που έχει στη διάθεσή της η Ευρωπαϊκή Ένωση μετά τη συνθήκη της Λισαβόνας. Δεν θα επικεντρωθούμε πολύ πάνω σε αυτά, απλώς κάτι θα αναφέρω γι' αυτό. Και το τέταρτο τμήμα είναι ίσως ένα από τα πιο σημαντικά, διότι κάνει συστάσεις όσον αφορά την πολιτική που πρέπει να ακολουθήσουμε. Τώρα, όπως ξέρετε, η Ρώμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι διαφορετική πληθυσμοί. Είναι πολύ δύσκολο να ετοιμάσουμε συμπεράσματα και συστάσεις που να ισχύουν για όλους, για όλες τις χώρες και για όλες τις ομάδες Ρώμα που είναι διασπαρμένες στις διάφορες ευρωπαϊκές χώρες. Σε ορισμένε χώρες είναι περιθωριοποιημένοι κατά πολύ, σε άλλες χώρες είναι περισσότερο ενταγμένοι στην κοινωνία. Ο κοινό παρονομαστής είναι ότι οι περισσότεροι βρίσκονται σε κατάσταση κοινωνικού αποκλεισμού, ένδυας και ανεργίας. Με χαμηλά επίπεδα κατάρτισης επίσης. Τώρα για να έχουμε μια ιδέα πρέπει να ξέρετε ότι πρόκειται για 10 με 12 εκατομμύρια ανθρώπους που σημαίνει ότι ο συνολικός του αριθμό είναι όσο ο πληθυσμός μιας χώρας όπως η Ουγγαρία ή η Ελλάδα. Συγκεντρώνονται κυρίως στην Ατινοτολική Ευρώπη, αλλά πάρα πολλοί από αυτούς βρίσκονται και στην Ισπανία. Η κατάσταση των Ρώμα έχει επιδεινωθεί επειδή υπήρξε αναδιάρθρωση των οικονομιών στην Ανατολική Ευρώπη και υπήρξε μια μεταβατική περίοδος. Οι πληθυσμοί των Ρώμα από τις χώρες αυτές έχουν μπει στο περιθώριο και συνεχίζουν να μπαίνουν στο περιθώριο όλο και περισσότερο. Γι' αυτό και η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται μια συνεκτική πολιτική ώστε να εντάξει τους Ρώμα μέσα στις ευρωπαϊκές κοινωνίες και να τους βοηθήσει να πετύχουν καλύτερα επίπεδα εκπαίδευσης και υγείας. Και αυτό δεν είναι προ δικό του όφελο μόνο, είναι και προ όφελο ολόκληρη τη Ευρώπη. Όπω έχει δείξει και η Παγκόσμια Τράπεζη πρόσφατα σε μια εκθεσή τη, κοστίζει χρήματα ο αποκλεισμό στον Ρώμα. Και πολλά μάλιστα στι ε, χώρε που εμπλέκονται στον αποκλεισμό αυτό. Η μελέτη που ετοιμάσαμε με τους συναδέρφους βασίζεται σε 12 διαφορετικές χώρες, όπως σας είπα και πριν. Αυτό που σας παρουσιάζουμε σήμερα είναι την συνθετική έκθεση όσον αφορά και τις 12 αυτές χώρες. Η έκθεση όμως δεν ξεκίνησε μέσα σε ένα κενό. Έχουν γίνει πολλές προσπάθειες σε πολιτικό επίπεδο τα τελευταία χρόνια από την Ευρωπαϊκή Ένωση υπέρ των Ρώμα, αλλά και από άλλους οργανισμούς. Όντως είναι πολλοί οργανισμοί οι οποίοι έχουν ασχοληθεί με θέματα που αφορούν τους Ρώμα. Πρώτα απ' όλα έχουμε βέβαια τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Συμβούλιο, Κομισιόν, επίσης το Συμβούλιο για την Υγεία και τους Καταναλωτές, όπως επίσης και Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Μετά τη Λισαβόνα, μάλιστα, το θέμα των θεμελιωδών δικαιωμάτων έχει αποκτήσει μεγαλύτερη σημασία. Και τι λένε τα θεμελιώδη δικαιώματα, ότι απαγορεύονται διακρίσεις. Και αυτό είναι πολύ βασικό όσον αφορά τους Ρώμα. Έπειτα η ΕΚΡΙ έχει ετοιμάσει πολλές ε, εκθέσεις τον τελευταίο καιρό από το Συμβούλιο της Ευρώπης και διάφορα δίκτυα που συμμετέχουν και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Υπάρχουν λοιπόν πολλέ εκθέσει. Το Συμβούλιο τη Ευρώπη, όπω σα είπα, μέσω τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, κατά του ρατσισμού και τη ε, αδιαλαξία. Και δίκτυα υπάρχουν σε πολλέ χώρε και σε διάφορα επίπεδα. Συμμετέχουν και εκπρόσωποι των ίδιων των Ρώμα. Είναι η Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα για την Ένταξη των Ρώμα υπό την αιγύδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έχουν γίνει διάφορες εσκέψεις κορυφής για τους Ρώμα, πρόσφατα μάλιστα. Υπάρχει το δίκτυο των Ρώμα, που είναι μια οργάνωση η οποία θέλει τα ωφέλη για τους Ρώμα να μεγιστοποιηθούν από πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συνεργάζεται με μια οργάνωση μη κυβερνητικών οργανώσεων τέλος υπάρχει και το Decade of Roma Inclusion που συμμετέχουν ε, διάφορες οργανώσεις και από τις 12 χώρες που μελετάμε και όπου συμμετέχουν πολλοί πολίτες Ρώμα. Στόχος της έκθεσής μας είναι να συγκεντρώσουμε τη γνώση μας και να ενημερωνόμαστε συνέχεια από τις μελέτες που κάνουμε στις διάφορες χώρες για να καταλήξουμε ποια είναι η πολιτική η οποία λειτουργεί καλύτερα και σε ποια χώρα. Έτσι θα δούμε τι πρέπει να κάνουν τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα τώρα που βρισκόμαστε στην εποχή μετά τη Λισαβόνα, ώστε να έχουμε τις βέλτιστες πρακτικές στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να χρησιμοποιούμε τα καλύτερα δυνατόν μέσα και να βελτιώσουμε την ζωή των πληθυσμών Ρώμα μέσα στην Ευρώπη. Αναγνωρίζουμε επίσης ότι η κατανομή των Ρώμα είναι άνηση μεταξύ των χωρών μελών αλλά και μέσα στα διάφορα κράτη-μέλη. Το θέμα αυτό της κατανομής, της εδαφικής κατανομής τους είναι πολύ σημαντικό. Ορισμένες καινούργιες χώρες μέλη έχουν ε, μεγάλα ποσοστά Ρώμα μεταξύ των πολιτών τους 7%, 5 με 7% σε ορισμένες χώρες όπως είναι η Ρουμανία, η Βουλγαρία. Και η Ισπανία όμως έχει ένα υψηλό ποσοστό Ρώμα. Που είναι όμως πολύ συγκεντρωμένη στην Ανταλουσία στην Ανδαλουσία, στην Νότια Ισπανία δηλαδή. Πολιτική ανάλυση. Συνολικά το νομικό πλαίσιο που διαθέτουν οι διάφορες χώρες διαφέρει από χώρα σε χώρα. Ορισμένες αναγνωρίζουν τους Ρώμα σαν μια χωριστή εθνική μειονότητα ή έχουν υιοθετήσει νομοθεσία όσον αφορά τους Ρώμα ως μειονότητα. Η Γερμανία, για παράδειγμα, η Ουγγαρία, η Πολωνία, η Ρουμανία και η Σλοβακία. Η Ισπανία έχει νομοθεσία για την κοινωνική ένταξη των Ρώμα και η Ουγγαρία αναγνωρίζει 13 εθνικές μειονότητες, μεταξύ των οποίων και τους Ρώμα. Η Πολωνία, απ' την άλλη, αναγνωρίζει τους ε, Ρώμα σαν εθνική μειονότητα στο Σύνταγμά της. Υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις επίσης Και η διαφοροποίηση αυτή, όσον αφορά την αναγνώριση των Ρώμα, διαφοροποιεί και τις πολιτικές αντιμετώπισης των προβλημάτων που προκύπτουν. Κάθε χώρα τώρα, πέρα από το ότι έχει διαφορετικά νομικά μέσα, έχει και διαφορετικά θεσμικά μέσα στη διάθεσή της. πρέπει να πούμε ότι οι διοικητικές δομές, οι θεσμικές δομές των ε, χωρών διαφέρουν και μεταξύ των χωρών μελών, αλλά και μεταξύ διαφορετικών κυβερνήσεων που περνάνε από κάθε χώρα. Στις καινούργιες χώρες κυρίως το πρόβλημα είναι μεγάλο. Έπρεπε για να ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι νέες χώρες να δείξουν ότι σέβονται τα δικαιώματα των μειονοτήτων. Σε ορισμένε νέες χώρες μέλη λοιπόν το θεσμικό πλαίσιο δεν είναι τόσο αναπτυγμένο όπως ήταν στις παλιότερες χώρες. Οπότε δυσκολεύονται να εφαρμόσουν μέτρα τα οποία προστατεύουν τους ε, Ρώμα. Παρόλα αυτά υπάρχει μια βάση πάνω στην οποία μπορούμε να χτίσουμε και να βελτιώσουμε την κατάσταση εφόσον η Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίξει τις διάφορες χώρες. Ένα ενδιαφέρον σημείο που έχει να κάνει με το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο είναι ότι σε αρκετές χώρες υπάρχουν διπουργικές επιτροπές οι οποίες συντονίζουν την πολιτική για τους Ρώμα. Υπάρχουν επικρίσεις βέβαια όσον αφορά την εφαρμογή, την έλλειψη εφαρμογής των ε, ρυθμίσεων. Συχνά το πρόβλημα είναι ο συντονισμός που είναι αδύναμος. Στην Τσεχία, για παράδειγμα, στην Ελλάδα υπάρχει η Διπουργική Επιτροπή για τους Ρώμα, υπάρχει ένα συμβούλιο για την ένταξη των Ρώμα στην Ουγγαρία, στη Σλοβακία υπάρχει μια υπηρεσία για να εξυπηρετεί τη κοινότητα των Ρώμα. Και τέλος στην Ισπανία υπάρχει ένα κρατικό συντονιστικό συμβούλιο. Αλλού την αρμοδιότητα την έχουν κάποια υπουργεία. Στη Βουλγαρία το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. Στην Πολωνία το τμήμα περιφερειών και εθνικών μειονοτήτων. Και στη Ρουμανία υπάρχει μια εθνική υπηρεσία που είναι αρμόδια για τους Ρώμα. Όσον αφορά την οργάνωση των κρατών, διαπιστώνουμε ότι ορισμένες χώρες επικεντρώνουν την πολιτική τους σε εθνικό επίπεδο. Άλλες ε, έχουν περιφερειακές ε, διαφορές. Δηλαδή βρίσκεται η διαχείριση του θέματος σε πιο χαμηλό επίπεδο. Υπάρχει αποκέντρωση των αρμοδιοτήτων, όπως στη Γερμανία που είναι ομοσπονδιακή, ή στην Ιταλία με τις περιφέρειες και τις επαρχίες, στην Ισπανία με τις αυτόνομες κοινότητες κλπ. Τώρα για τους διάφορους τομείς πολιτικής. Σας είπα ότι κυρίως εδώ πρόκειται για την εκπαίδευση και την απασχόληση. Η εκπαίδευση. Είναι πολύ σημαντικό στοιχείο για να διευκολυνθεί η κοινωνική ένταξη των Ρώμα. Ο αποκλεισμό από την εκπαίδευση δημιουργεί έναν φαύλο κύκλο και βάζει στο περιθώριο τους Ρώμα από πολύ μικρή ηλικία ήδη. Γι' αυτό είναι πολύ βασικό να υπάρχουν πολιτικά μέτρα που να διευκολύνουν την εκπαίδευση και την κατάρτιση των πληθυσμών αυτών. Πρέπει να ενισχυθεί η δυνατότητα των ανθρώπων αυτών να πηγαίνουν στο σχολείο. Η χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το σκοπό αυτό πρέπει να είναι πολύ συγκεκριμένη, ώστε όντως τα παιδιά των Ρώμα να πηγαίνουν στο σχολείο και να παραμένουν στο σχολείο μέχρι να τελειώσει η υποχρεωτική εκπαίδευση, αντί να τον καταλείπουν ε, πολύ γρήγορα. Είναι πολύ βασικό αυτό, γιατί αποτελεί τη βάση πάνω στην οποία ε, μπορούν να δουλέψουν οι Ρώμα για να ενταχθούν αργότερα στην ε, κοινωνία, στην αγορά εργασίας κλπ. κλπ. Αλλιώς είναι ένας φαύλος κύκλος. Οι Ρώμα δεν συμπληρώνουν ε, τον εκπαιδευτικό κύκλο, πράγμα το οποίο τους βάζει στο περιθώριο όσον αφορά την αγορά εργασίας, με εξαίρεση την Ισπανία, η οποία βελτιώνει την ένταξη των Ρώμα στην εκπαίδευση από πολύ νωρίς. Οι διάφορες χώρες ακολουθούν διαφορετικά σχέδια, διαφορετική στρατηγική, όπως είπαμε και πριν. Και φαίνεται αυτό από τον πίνακα όπου αναφέρονται διάφορες χώρες. Πάντως, υπάρχει ένα ευρύ φάσμα μηχανισμών και μέτρων που χρησιμοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το πρόβλημα είναι ότι το καθένα από αυτά τα μέτρα είναι ένα μόνο μέρος Δηλαδή, αν δείτε συνολικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση τι ισχύει, θα δείτε ότι το φάσμα είναι ευρύ. Υπάρχουν πάρα πολλές πρωτοβουλίες που θα μπορούσαν ε, να αποτελέσουν ε, παράδειγμα για άλλες χώρες. Θα μπορούσαν δηλαδή να παραδειγματιστούν κάποιες χώρες από κάποιες άλλες και να χρησιμοποιήσουν τις καλύτερες δυνατόν πρακτικές. Πρώτα απ' όλα, πρόσβαση. Πρέπει τα παιδιά των Ρώμα να έχουν πρόσβαση στο εκπαιδευτικό σύστημα και να έχουν και κίνητρα βέβαια για να πάνε και να μείνουν στο σύστημα αυτό. Δεύτερον, κάτι άλλο σημαντικό είναι η βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης. Το εκπαιδευτικό σύστημα πρέπει να ανταποκρίνεται στις ειδικέ ανάγκες που έχουν οι Ρώμα. Τέτοια παραδείγματα έχουμε σε διάφορες χώρες με μεσολαβητές που χρησιμοποιούνται για να αποτελέσουν τον σύνδεσμο ανάμεσα στις οικογένειες και τα σχολεία, ώστε να βοηθήσουν τα παιδιά να ξεκινήσουν, να τους δίνουν κίνητρα για να παραμείνουν στο σχολείο και πολλές χώρες δίνουν τέτοια κίνητρα στις οικογένειες για να στέλνουν τα παιδιά τους στο σχολείο. Για την ε, βελτίωση της ποιότητας τι κάνουν οι διάφορες χώρες. Για παράδειγμα, καταρτίζουν κατάλληλα τους εκπαιδευτικούς, ώστε να μπορούν να αντιμετωπίσουν την ειδική ομάδα των Ρώμα. Υπάρχει, είπαμε, ένα ευρύ φάσμα μηχανισμών που αφαρμόζονται. Γιατί όμως δεν δίνουν και αποτελέσματα. Οι κύριες δυσκολίες εντοπίζονται στον θεσμικό συντονισμό ή στο ότι διοικητικά οι διάφορες χώρες ή σε τοπικό επίπεδο δεν υπάρχουν αρκετές δυνατότητες, υπάρχουν λίγοι πόροι ή δεν ε, υπάρχουν αρκετά κίνητρα, δεν δεσμεύονται οι αρμόδιοι αρκετά ή η χρηματοδότηση δεν είναι επαρκής, τελειώνει κάποια στιγμή και μετά τελείωσε και η κατάρτιση των Ρώμα. Τέλος, ε, έχουμε διαπιστώσει την απουσία του ελέγχου και της αξιολόγησης. Γιατί αν μια πολιτική που εφαρμόζεται δεν αξιολογείται, δεν ξέρουμε κατά πόσο είναι καλή, αν φέρνει αποτελέσματα ή όχι. Καλό θα ήταν λοιπόν να συμπεριλάβουμε και την αξιολόγηση. Εμείς από τη μελέτη μας διαπιστώσαμε ότι συχνά κανείς δεν ξέρει τι γίνεται και πόσο αποτελεσματικές είναι οι πρωτοβουλίες που λαμβάνονται. Χρειάζεται λοιπόν περισσότερη δουλειά σε αυτόν τον τομέα για να εντοπίζουμε τις καλύτερες πρακτικές. Ποσοτικά στοιχεία δεν μπορέσαμε να βρούμε για να αξιολογήσουμε τις προσπάθειες. Παρά το γεγονός λοιπόν ότι δεν υπάρχουν μελέτες αξιολόγησης, έχουν γίνει κάποιες προσπάθειες να αξιολογηθεί η επιτυχία ορισμένων πρωτοβουλειών. Και πρέπει για τελειώς, πώς να ξεκινήσει κανείς την διαδικασία ένταξης των παιδιών των Ρώμα στο εκπαιδευτικό σύστημα αν δεν έχει αξιολογήσει το σύστημα. Επειδή είναι πολύ συχνά στο περιθώριο Ρώμα, η προσχολική εκπαίδευση έχει τεράστια σημασία. Έπειτα πρέπει να υπάρχουν και δεύτερες ευκαιρίες για παιδιά που δυσκολεύονται μέσα στο εκπαιδευτικό σύστημα, είτε λόγω οικονομικών δυσκολιών, είτε επειδή αντιμετωπίζουν ε, διακριτική μεταχείριση σε βάρος τους. Εκεί πρέπει να υπάρχει μια παραπάνω προσπάθεια και μια παραπάνω ευκαιρία που δίνεται στα παιδιά αυτά. θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε την εμπειρία ορισμένων χωρών και να χτίσουμε πάνω σε αυτήν. Έπειτα είναι σημαντικό να υπάρχουν και κάποιοι έλεγχοι με τα αποτελέσματα των ε, παιδιών στην εκπαίδευση. Τώρα, σύντομα θα σας μιλήσω για την ε, απασχόληση επίσης. Υπάρχουν πολλά μέτρα που εφαρμόζονται όσον αφορά την απασχόληση. Πολλές κυβερνήσεις έχουν προσπαθήσει ξανά και ξανά να αναλάβουν πρωτοβουλίες στον ε, τομέα αυτό, αλλά οι προσπάθειες ήταν πάντα σποραδικές και ποτέ δεν υπήρξε συνέχεια. Είτε πρόκειται για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης για του Ρώμα, είτε υπήρχε ειδική πολιτική στην αγορά εργασίας υπέρ των Ρώμα, είτε πρόκειται για προγράμματα κατάρτισης στο Ρώμα, είτε κάτι άλλο πολύ σημαντικό, ακριβώς επειδή υπάρχει διακριτική μεταχείριση σε βάρος στο Ρώμα, υπήρξαν συχνά προγράμματα για να βοηθήσουν τα κράτη του Ρώμα να φτιάξουν τις δικές τους επιχειρήσεις. Ή και στη... και στη Γεωργία ε, μικρές επιχειρήσεις, συνεταιρισμοί, η Ρώμα έχουν την ευκαιρία να δουλέψουν τη γη. Τα προβλήματα μερικές φορές είναι πολύ συγκεντρωμένα γεωγραφικά. Δηλαδή, σε ορισμένες περιοχές βρίσκονται σε ιδιαίτερα δυσμένη κατάσταση η Ρώμα. Πολλές φορές σε δύσκολες αγροτικές περιοχές. Το τελευταίο μέτρο που έχουμε εντοπίσει είναι η προσπάθεια που γίνεται από να προσφέρουν ε, στους Ρώμα την ικανότητα να διαχειριστούν ήδη τη ζωή τους. Υπάρχουν συχνά προβλήματα με την εφαρμογή των μέτρων. Υπάρχουν προγράμματα δράσης σε εθνικό <coughs> επίπεδο για την απασχόληση. Τα μέτρα για την άμεση πρόσληψη των Ρώμα διαπιστώσαμε επίσης ότι δεν απέδωσαν πολύ. Οι διοικητικές διαδικασίες από την άλλη μεριά για να φτιάξουν οι Ρώμα τη δική τους επιχείρηση είναι ιδιαίτερα γραφειοκρατικές και δυσκολεύουν την πρόσβαση των Ρώμα. Εδώ βλέπετε την τελευταία μου διαφάνεια για τις βέλτιστες πρακτικές όσον αφορά την απασχάληση απασχόληση. Ίσως να έχετε υπόψη σας, πολλοί από εσά, τα προγράμματα Αξεντέρ, που είναι βοήθεια στους Ρώμα από κέντρα που υπάρχουν ειδικά για αυτούς σε διάφορες πόλεις και τους προσφέρουν προγράμματα κατάρτισης και βοήθεια για να βρουν κάποια δουλειά ή να φτιάξουν τη δικιά τους επιχείρηση. Πολλές χιλιάδες από τους Ρώμα στη στην Ισπανία έχουν βοηθηθεί από τέτοιου είδου προγράμματα. Στην Ουγγαρία υπάρχει κάτι αντίστοιχο που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο με καλά αποτελέσματα. Είναι πάλι μια ολοκληρωμένη προσέγγιση που φαίνεται ότι στέφεται από επιτυχία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Αυτό πρώτο μέρος της συζήτησης θα το ακολουθήσει ένα δεύτερο μέρος και προτείνω να είμαστε πιο σύντομοι, διότι έχουμε μόνο μία ώρα και ένα τέταρτο για τη συζήτηση. Και επίσης θα θέλαμε και μία ενημέρωση από την συγγήτριά μα, την κυρία Ντερόκα, και γι' αυτό σας παρακαλώ θερμά να είσαστε πιο σύντομοι για να έχουμε, μπορούμε να ολοκληρώσουμε και το δεύτερο γύρο της συζήτησης. Ευχαριστώ. Όντως, θα προσπαθήσω να είμαι σύντομη. Αυτό το οποίο έχω σκοπό να παρουσιάσω είναι σύντομα τις βασικές μας ε, συστάσεις για την ακολουθητέα πολιτική. Είναι το πρώτο σχέδιο αυτό συστάσεων. Είναι λοιπόν ενδεικτικές οι προτάσεις αυτές και όχι οριστικές ε, ως αποτέλεσμα της μελέτης που έχουμε κάνει. Λοιπόν, οι συστάσεις μας για την πολιτική επί του θέματος στηρίζονται σε τέσσερις ε, πυλώνες. Καταρχάς πρέπει να συγκεκριμενοποιήσουμε την προσέγγιση μας. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, να είμαστε σαφείς, γιατί εξ αρχής πρέπει να μπορέσουμε να ε, χαράξουμε μία συνεπή και συνεκτική πολιτική. Δεύτερον, ο δεύτερος πυλώνας είναι η βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των θεσμικών ε, οργάνων ο τρίτος πυλώνας είναι η βελτίωση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας ε, της πολιτικής επί τη βάση αξιολογήσεων ε, των προγραμμάτων που ισχύουν και το τέταρτο είναι η διατύπωση συγκεκριμένων συστάσεων. Επανέρχομαι στον πρώτο πυλώνα. Ποια είναι η βασική μας προσέγγιση. Ε, τι προτείνουμε μέσα σε ποιο πλαίσιο. Ποια είναι η προσέγγιση μας την οποία το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, έχει ήδη χαρακτηρίσει ως συνεκτική. Μία πολιτική που ε, ταυτίζεται με την συνοχή και με την συνέχεια αυτό που θέλουμε να εδραιώσουμε είναι να έχουμε σωστές ε, σχέσεις με όλους τους εμπλεκόμενους ε, φορείς που ε, μέσα στο πλαίσιο των οποίων εμπίπτει το θέμα της ενσωμάτωσης των Ρώμα. Ο πρώτος τέτοιος πυλώνας, η πρώτη αυτή λοιπόν πολιτική, περιλαμβάνει την ισότιμη πρόσβαση των παιδιών των Ρώμα στην παιδεία, στις ευκαιρίες μόρφωσης, εκπαίδευσης. Αυτή είναι μία προσέγγιση, μία στρατηγική μακροχρόνια. Ε, είναι η πρώτη μας προτεραιότητα, απόλυτη προτεραιότητα. Διότι η επίπτωση μιας τέτοιας στρατηγικής ε, θα είναι πρόθεσμη και μακροπρόθεσμη βεβαίως. Η δεύτερη μας προσέγγιση επικεντρώνεται στην συγκέντρωση επαρκών στοιχείων, ε, κονδυλίων συγγνώμη, για να διευκολύνουμε την πρόσβαση των Ρώμα στην αγορά εργασίας. Πρέπει λοιπόν να μπορέσουμε να βοηθήσουμε και σε αυτό τον τομέα. Η τρίτη, ο τρίτος τομέας αυτού του πρώτου πυλώνα είναι η κοινωνική ζωή, η ενσωμάτωση στην κοινωνική ζωή, η κάλυψη από τους οργανισμούς ε, κοινωνικής ασφάλειας, η παροχή υπηρεσιών φροντίδας των παιδιών, ε, φροντίδας ε, υγείας και όλα τα συναφή κοινωνικά μέτρα για τη βελτίωση των συνθήκων ζωής. Οι τέσσερις πυλώνες λοιπόν αυτοί υπάρχουν ήδη διότι ήδη η Ευρωπαϊκή Κομισιόν ε, και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με τη βοήθεια του Διευθυντικού Ταμείου έχουν επισημάνει ακριβώς ε, τις ανάγκες αυτές που, στις οποίες πρέπει να δώσουμε προτεραιότητα μέσω της περιφερειακής πολιτικής. Η περιφερειακή πολιτική και το περιφερειακό ταμείο είναι πολύ σημαντικά διότι, διότι έτσι μπορούμε να εφαρμόσουμε οριζόντια μέτρα σε διατομεακές πολιτικές διότι πρέπει ταυτόχρονα να αντιμετωπίσουμε την πρόσβαση στην παιδεία, το οικονομικό πρόβλημα, την κοινωνική και πολιτιστική ενσωμάτωση της συνθήκες διαβίωσης κλπ. Άρα λοιπόν και η περιφερειακή πολιτική αλλά και η τοπική αυτοδιοίκηση είναι σημαντική μοχλή που θα βοηθήσουν την ενσωμάτωση των Ρώμα. Εδώ βλέπετε ένα γράφημα που δείχνει τις διάφορες, τη σύνδεση μεταξύ των διαφόρων τομέων και πολιτικών ε, και τις ε, διάφορες πτυχές της ενσωμάτωσης τις οποίες πρέπει να ε, εστιάσουμε την προσοχή μας η κοινωνική πολιτική, η εργασιακή πολιτική και τους υποτομείς. Είναι οι πρωτογενείς και δευτερογενείς τομείς της ενσωμάτωσης, τους οποίους θέλουμε να προωθήσουμε και οι διασυνδέσεις μεταξύ τους. Αυτή είναι μια θεωρητική προσέγγιση βέβαια και το πρόβλημα και η περιπλοκότητα του προβλήματος είναι πολύ μεγάλη, διότι εδώ πρέπει να χαράξουμε μια στρατηγική που να μπορέσει να τα προωθήσει όλα αυτά με συνεκτικό τρόπο. Καταρχάς, λοιπόν, όσο αφορά το στόχο βελτίωσης ε, των, ε, της ζωής των Ρωμά. Καταρχάς, η ανάπτυξη των, ε, του θεσμικού δυναμικού Αυτό καλύπτει τους τομείς της ε, στέγασης, διαβίωσης και παιδείας και την εφαρμογή των βέλτιστων πρακτικών, συγκριτικών πολιτικών, ανταλλαγής πληροφοριών. Αυτό μπορεί να αποτελέσει ένα θαυμάσιο κανάλι για την ανταλλαγή εμπειριών και από τις δύο πλευρές όσον αφορά την προηγούμενη εμπειρία, τις βέλτιστες πρακτικές ε, για τη βελτίωση όλων αυτών των, των, των θεμάτων. Η δεύτερη πτυχή, ο δεύτερος τομέας δράσης που έχουμε επισημάνει στη μελέτη μας είναι η υιοθέτηση συστηματικής παρακολούθησης και αξιολόγησης. Σας είπα ήδη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ελευθερωτικό Ταμείο και άλλοι φορείς εμπλέκονται σε όλη αυτή την προσπάθεια. Αλλά στις διάφορες εθνικές εκθέσεις βλέπουμε ότι πάρα πολλές ε, αναφορές αξιολόγησης και παρακολούθησης λείπουν. Δεν υποβάλλονται λοιπόν στα πλαίσια των εθνικών εξέσεων. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχει μια ανεπάρκεια παρακολούθησης και αξιολόγησης στα πλαίσια των εθνικών πολιτικών. Πρέπει λοιπόν οπωσδήποτε για να μπορέσουμε να αξιολογήσουμε το ποιοτικό και ποσοτικό χαρακτήρα των μέτρων, να έχουμε μία έκθεση αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας των πολιτικών για να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε μία συστηματική προσέγγιση της ενσωμάτωση των Ρώμα. Επίσης, μέσα στα πλαίσια της εποπτείας και αξιολόγησης, πρέπει οπωσδήποτε να καθορίσουμε ποιος θα κάνει τι. Δηλαδή, πού θα ανασέσουμε αυτές τις εξαίσεις αξιολόγησης. Έχουμε εξωτερικούς σύμβουλους και εσωτερικές υπηρεσίες που μπορούν να το κάνουν. Αυτό που είναι σημαντικό είναι να τονίσουμε την εσωτερική αξιολόγηση. Αυτή θα πρέπει να ακολουθήσει μία ε, συμμετοχική διαδικασία, διότι θέλουμε να λάβουν μέρος σε αυτή την αξιολόγηση και εκπρόσωποι των ε, Ρωμά ε, που δρούν επιτόπου και ξέρουν τις επιτόπιες συνθήκες. Γι' αυτό πρέπει να έχουμε μια συγκεκριμένη τεχνική αξιολόγηση και αυτή η τεχνική θα πρέπει να καλύπτει οπωσδήποτε και την άμεση συμμετοχή των Ρώμα στις δραστηριότητες. Έτσι και μόνον έτσι θα μπορέσουμε να αυξήσουμε τη βούληση των Ρωμά να συμμετάσχουν στις επιτυχές, στα επιτυχή αυτά προγράμματα. Να συμμετάσχουν έτσι ώστε τα προγράμματα τελικά να είναι αποτελεσματικά και επιτυχή. Αυτή λοιπόν ε, είναι η εσωτερική διαδικασία. Τώρα, η εξωτερική εμπειρογνωμοσύνη σε εθνικό και τοπικό επίπεδο είναι επίσης πολύ σημαντική, διότι εδώ μέσω των θεσμικών οργάνων πρέπει να ξέρουμε πόσο έχει προχωρήσει το πρόγραμμα, αν έχει προχωρήσει και πόσο έχει επιτύχει ή όχι, για να αποφύγουμε επικαλύψεις και λάθη που έχουν γίνει στο παρελθόν. Και πολύ σύντομα Βλέπετε εδώ την ανοιχτή μέθοδο συντονισμού και αξιολόγησης που ακολουθούμε, ε, ε, αξιολογώντας την αποτελεσματικότητα των πολιτικών. Και ε, τώρα θα έρθω στο θέμα της βελτίωσης των θεσμικών, της θεσμικής συνεργασίας, του θεσμικού συντονισμού. Δηλαδή πώς μπορούμε στο ευρωπαϊκό επίπεδο να συντονίσουμε όλους αυτούς τους φορείς και όλες αυτές τις διευθύνσεις μέσα στο ευρωπαϊκό επίπεδο που ασχολούνται με αυτό το θέμα. Συντονισμός λοιπόν και συνεργασία. Θέλουμε με πιο συνεκτικό τρόπο να συντονίσουμε τις διάφορες τομεακές και διακλαδικές δράσεις που αφορούν τους Ρώμα. Το δεύτερο δεύτερο, η δεύτερη πρόταση είναι η βελτίωση της, του συντονισμού σε εθνικό επίπεδο. Στην έκθεση των 12 χωρών διαπιστώσαμε ότι υπάρχει μια πάρα πολύ τεμαχισμένη, διάσπαρτη και μη συντονισμένη εμπειρία στο θέμα της αντιμετώπισης των Ρώμα και πρέπει οπωσδήποτε να βελτιώσουμε το συντονισμό για να εξοικονομήσουμε πόρους και να αυξήσουμε την αποδοτικότητα. Υπάρχει λοιπόν κατατεμαχισμός δράσεων και προσπαθειών και αυτό πρέπει να, εδώ πρέπει να εφαρμόσουμε έναν ε, συντονισμό. Επίσης, στο διεθνές επίπεδο πρέπει να επιτύχουμε στενότερο συντονισμό και συνεργασία, ώστε να συνεργαστούμε πιο στενά με τους διεθνείς οργανισμούς, όπως η Παγκόσμια Τράπεζα, το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΟΗΕ, το Διεθνή Γραφείο Εργασίας, όλους λοιπόν τους διεθνούς φορείς μέσα στους οποίους ε, οι οποίοι και αυτοί έχουν μέτρα ή προγράμματα για τους Ρώμα. Όλα αυτά πρέπει να συντονιστούν καλύτερα. Και βεβαίως πρέπει να ε, βελτιώσουμε και την ευρωπαϊκή, το ευρωπαϊκό δυναμικό επιχειρηματικής δράσης. Δηλαδή πρέπει να δημιουργήσουμε ένα φορέα συντονισμού, μια υπηρεσία, μια επιτροπή για να ενισχύσει όλους αυτούς που συμμετέχουν σε αυτό το πρόγραμμα. Όπως παραδείγματο χάρη μια ευρωπαϊκή πλατφόρμα για τους Ρώμα. Μπορεί να είναι μια επιτροπή, μπορεί να είναι εν πάση περιπτώσει ένας ευρωπαϊκός φορέας που θα παρακολουθεί και θα βοηθήσει τον καλύτερο συντονισμό της στρατηγικής και όλων των συναφών πολιτικών and um, Οπότε, προχωρώ πολύ γρήγορα στο θέμα της παιδείας, το οποίο ήδη έχω θίξει. Βασικός στόχος είναι η βελτίωση της πρόσβασης, η ποιοτική βελτίωση, η μόρφωση και ε, ε, συμπερίληψη ε, των γυναικών Ρώμα, δηλαδή το θέμα της φιλετικής, της διάστασης του φύλου, να ενισχυθεί και επίσης η ανάπτυξη ε, τεχνολογίας, σύγχρονης τεχνολογίας, ε, ε, μάθησης εξ αποστάσεως, διαβίου μάθησης ε, και ε, τέλος πάντων κάλυψη όλων των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και συμμετοχή των Ρώμα. Απασχόληση και συμμετοχή στην αγορά εργασίας. Εδώ θέλουμε να εφαρμόσουμε άμεσα μέτρα για μόνιμη και προσωρινή ημερική απασχόληση, επίσης ε, πολιτικές ε, στην αγορά εργασίας, να τους δώσουμε τη δυνατότητα να ξεκινήσουν μικρές επιχειρήσεις, ατομικές επιχειρήσεις, να εφαρμοστούν μέτρα σε τοπικό επίπεδο, μέσω τοπικής αυτοδιοίκησης, επίσης στην Ήπεθρο. Στην Ήπεθρο, σε υπαίθριες και ε, αγροτικές περιοχές, τα θέματα, τα προβλήματα είναι οξία και πρέπει και εκεί να βοηθήσουμε για να, δημιουργηθούν, να δημιουργηθεί απασχόληση. Ε, επίσης να βελτιώσουμε το δυναμικό, τη δυνατότητα δραστηριότητας ε, των γραφείων εργασίας, δηλαδή των αντίστοιχων ΟΑΕΔ και κρατικών υπηρεσιών ε, και επίσης να βελτιώσουμε τη διάσταση του φύλου σε όλα τα θέματα. Ε, στέγαση, να βελτιώσουμε τις, ε, τις συνθήκες διαβίωσης εκεί όπου ζουν οι Ρώμα, σε αστικές και υπαίθριες περιοχές, παροχή των βασικών υποδομών, και επίσης ένα χωροταξικό πρόγραμμα. Αυτό είναι πάρα πολύ ευαίσθητο διότι οι τοπικοί δήμοι και κοινότητες πρέπει να κάνουν μεγαλύτερες προσπάθειες για να παράσχουν τις βασικές ευκολίες στέγας και διαμονής στον Ρώμα. Η προσφορά σπιτιών, η πρέπει να ε, αυξηθεί. Πρέπει να δημιουργήσουμε περισσότερες εργατικές κατοικίες, αν θέλετε, για να μπορέσουμε να στεγάσουμε τους Ρώμα. Είναι ένα πάρα πολύ περίπλοκο θέμα, διότι εμπλέκονται και οι τοπικές αυτοδιοικήσεις και δεν έχουμε τον καιρό τώρα να τα μελετήσουμε όλα. Θα έλεγα, λέει ο Πρόεδρος, να μας παρουσιάσετε τις συστάσεις σας. Ε, άλλες διάφορες πρωτοβουλίες στην υγεία, και στα δημοσιονομικά μέσα, ε, χρηματοδοτικά μέσα, μέσω του διαφορετικού ταμείου, του Ταμείου Συνεχής του Αγροτικού και Ταμείου για την Ανάπτυξη της Υπέθρου και Κοινωνικών Προγραμμάτων, θέλουμε να βελτιώσουμε τη χρηματοδότηση. Το, όλα αυτά τα ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να προσαρμόσουν τις πολιτικές τους για να ενσωματώσουν την πολιτική των Ρώμα και ανακαλύψουν τις απαραίτητες ανάγκες. Και καταλήγοντας θα αναφερθώ σε δύο βασικά θέματα που είναι οριζόντια. Καταρχάς το θέμα της συλλογής στοιχείων, της συλλογής δεδομένων είναι λίγα σημαντικό πρέπει να ξέρουμε ακριβώς για πόσους ανθρώπους μιλάμε, από απόψεως δημογραφικών δηλαδή δεδομένων πρέπει να συλλέξουμε τα απαραίτητα στοιχεία για να τα δώσουμε στους ηθήνοντες της πολιτικής για να έχουν τις κατάλληλες πληροφορίες στα χέρια τους για να συντάξουν τις τις πολιτικές. Επίσης, πρέπει κατά δεύτερο λόγο, εν κατακλείδη, να δημιουργήσουμε εκστρατείες ε, ενημέρωσης του κοινού ε, για την προβολή των, της πολιτιστικής διάστασης των Ρώμα ε, και για να γίνει το κοινό, να ευαισθητοποιήσουμε το κοινό ως προς αυτούς. Σας ευχαριστώ που τα είπα τόσο τηλεγραφικά λόγω πίεσης χρόνου. Ευχαριστώ πάρα πολύ και σας ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί βιαστήκατε. Τι να κάνουμε στην Επιτροπή μας, ε, το πρόγραμμα είναι ιδιαίτερα βεβαρημένο και σήμερα ε, έχουμε πολλά πράγματα και πρέπει να βιαστούμε. Καταρχάς να ακούσουμε από την εισηγήτρια να μας πει κάποιες πληροφορίες και έχω και έναν κατάλογο των μελών που θα ήθελα να πάρουν το λόγο. Θα ήθελα να σας ζητήσω να είστε σύντομοι, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο. Θα κλείσω εδώ τον κατάλογο. Δεν νομίζω ότι θέλει κανείς άλλος. Α, κάποιοι θέλουν ε, να προσθεθούν στον κατάλογο. Η κυρία Αλφάνο, η κυρία Ματιέ. Λοιπόν, ο κατάλογος έκλεισε. Και θα ακούσουμε τώρα την κυρία Γιαρόκα. Ευχαριστώ πάρα πολύ ε, κύριε Πρόεδρε, τα, δι, τα τρία πρώτα σχόλια θα αφορούν αφορούν την έκθεση. Και μετά, όταν ξεκινήσουμε την ανταλλαγή απόψεων, θα κάνω και άλλα τρία σχόλια. Για την έρευνα και τη μελέτη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσπάθεια, για τα πορίσματά σας. Ε, περιμένουμε με ενδιαφέρον να διαβάσουμε όλα τα πορίσματα. Και αυτό το οποίο ήθελα να τονίσω όσον αφορά τα ενδιάμεσα συμπεράσματα είναι ότι αυτό το οποίο θα έπρεπε να καταλάβει αυτή η Επιτροπή, και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, είναι ότι δεν θα πρέπει να μπορείτε να δείτε μόνο αυτά τα, οποία, αυτά τα μέτρα τα οποία ήδη υπάρχουν και αφορούν τους Ρώμα, π.χ. οδηγίες, αλλά θα θέλαμε να ξέρουμε για όλα τα κοινοτικά εργαλεία ή όργανα τα οποία μπορεί να είναι διαθέσιμα για τη στρατηγική μας. Μας είπατε για, την, το τρίτο τμήμα αυτού της έκθεσης. Για μας ε, οι συστάσεις είναι οι πιο σημαντικές. Γι' αυτό αυτό θέλουμε να καταλάβουμε. Αυτό είναι κάπου λίγο θεωρητικό. Θέλουμε να ξέρουμε σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία ποια είναι τα εργαλεία τα οποία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Το δεύτερο θέμα το οποίο ήθελα να θίξω, ε, χαίρομαι γιατί όλες αυτές, όλες αυτές οι εθνικές εκθέσεις είχαν κάποια κοινά στοιχεία, αλλά αυτοί οι ελάχιστοι κοινοί παρινόμαστές θα πρέπει να συγκεκριμενοποιηθούν, θα πρέπει να τους δούμε και να δούμε πώς μπορούμε να τους χρησιμοποιήσουμε σε ε, κοινοτικό επίπεδο μέσα στα πλαίσια της προσπάθειας συντονισμού αυτό είναι κάτι ενδιαφέρον. Επίσης, ε, για τη μελέτη της 15ης ε, Νοεμβρίου θέλουμε μια συγκεκριμένη σύσταση ή συγκεκριμένες συστάσεις ε, και όσον αφορά τη δομή αλλά και την σταδιακή ανάπτυξη της ε, κοινωτικής στρατηγικής. Πώς αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να εναρμονιστούν οι διάφορες δράσεις αλλά και τις ικανότητες που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή. Αυτά τα πράγματα θέλουμε να μάθουμε και γι' αυτό ζητήσαμε την μελέτη αυτή. Επιτρέψτε μου κύριε Πρόεδρε, η κυρία Πρόεδρε μάλλον, στη συγκεκριμένη στιγμή, να να προχωρήσω στα σχόλια που θέλω να κάνω τώρα ή να προχωρήσω μετά. Τι, τι θέλω εγώ σαν εισηγητής. Έχουμε 20 λεπτά στη διάθεσή μας. Έχουμε 10 ε, μέλη στον κατάλογο. Λοιπόν, ένα λεπτό. Ένα λεπτό έχει ο καθένας, αν μπορείτε και μετά θα ήθελα να σας ζητήσω να απαντήσετε ή να σκεφτείτε τις ερωτήσεις ε, που θα ακουστούν. Λοιπόν, σε ένα λεπτό. Λοιπόν, με τη μελέτη, με τα αποτελέσματα της μελέτης, αυτά ήταν τα σχόλια που ήθελα να κάνω σαν εισηγήτρια και απλώς προσβλέπω με ενδιαφέρον ε, τα συμπεράσματά σας. Ε, τώρα, σαν εισηγήτρια ήθελα να πω ότι αυτό το έγγραφο εργασία το οποίο έχουμε μπροστά μας και είναι πρόκειται για τη δεύτερη ανταλλαγή απόψεων ε, αφορά την πολιτική των Ρώμα και τη συγκεκριμένη νομική βάση που πρέπει να χρησιμοποιήσουμε. Και στο έγγραφό μου ήδη αναφέρω ότι αυτό το οποίο θέλουμε να εξετάσουμε τώρα είναι το πλαίσιο και η δομή της συνεργασίας πώς τα κράτη-μέλη, τα θεσμικά όργανα της κοινότητας, οι ενδιαφερόμενοι πλατφόρμες των Ρώμα, η Task Force, πώς οι διάφορες επιτροπές μπορούν να συνεισφέρουν σε αυτό το πλαίσιο. Δεύτερον, πέραν αυτού του βασικού μηνύματος ότι θέλουμε δηλαδή μια κοινή ευρωπαϊκή στρατογική, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ποιες είναι οι συνέπειες όλες τις πολιτικές και θα πρέπει η Ευρώπη να καταλάβει ότι μόνο με ε, νομικά δεσμευτικά κείμενα μπορούμε να πετύχουμε το στόχο μας. Το είπατε κι εσείς αυτό ότι χρειάζεται, δεν ε, συμβαίνει πάντα βέβαια. Αυτά ζητάμε και επειδή είναι κρίσιμη στιγμή, επαναλαμβάνουμε τα αιτήματά μας, ε, γιατί η Κομισιόν σε λίγους μήνες θα υποβάλει προτάσεις για αυτές τις στρατηγικές. Ξέρουμε ότι η Ουγγρική Προεδρία είναι έτοιμη να αναλάβει τις συστάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, επομένως είναι πολύ σημαντικό για όλους μας να ενδυναμώσουμε αυτό το μήνυμά μας, ότι εδώ και έξι χρόνια είμαστε ενωμένοι, ότι χρειαζόμαστε μια στρατηγική για τους Ρωμά και όπως είπα και την προηγούμενη φορά, τα τέσσερα πιο σημαντικά στοιχεία τα οποία αφορούν τις ε, κοινωνικο-οικονομική ε, κατάσταση, αφορούν την, ε, τη διακριτική μεταφορά την, ε, το ότι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ε, και την, ε, τον περιφερειακό χαρακτήρα αυτής του, αυτού του αποκλεισμού και θα πρέπει να βρούμε μία απάντηση σε αυτά τα στοιχεία τα οποία ανέφερα και αν βρούμε αυτή την απάντηση τότε θα έχουμε μία αποτελεσματική στρατηγική για τους Ρωμά. Θα ήθελα να ακούσω τα σχόλια όλων γιατί θα πρέπει να δώσουμε ένα σαφές μήνυμα στην προεδρία, ε, την επερχόμενη προεδρία της Ουγγαρίας, η οποία θέλει ακριβώς να τα λάβει υπόψη της. Καλό θα λέει η πρόεδρος να ακούσουμε και τα άλλα μέλη. Η Ρενάτα Βέμπερ είναι η επόμενη ομιλήτρια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρέπει να σας πω ότι η μελέτη είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Πρέπει να σας πω όμως ότι εστιάζεται αποκλειστικά στις κοινωνικο-οικονομικές πτυχές και αυτή είναι μία ε, μελέτη την οποία ζητήσαμε εμείς και όχι η Επιτροπή Απασχόλησης. Ε, και ήλπιζα και περίμενα ότι, και περιμένω τουλάχιστον ότι οι συγγραφείς θα επαναπροσανατολίσουν την μελέτη και να υπάρχουν και θέματα διακριτικής μεταχείρισης, ε, αποκλεισμού, πολιτικών ελευθεριών, θέματα δηλαδή που μας αφορούν και θα έπρεπε να αναφέρονται στην έκθεση αυτή. Γιατί θα πρέπει και στην έκθεση τη εισηγήτριας να υπάρχουν όλα αυτά τα στοιχεία. Εάν θέλουμε να βοηθήσουμε την Επιτροπή την, στην προσπάθειά της να προτείνει μια συγκεκριμένη στρατηγική, τότε θα πρέπει να στείλουμε ένα σαφές μήνυμα. Και νομίζω ότι μπορεί να είναι διαπολιτικό, αν θέλετε, διακομματικό το μήνυμα και όχι για όλα τα θέματα, συγγνώμη, για όλες τις πτυχές. Όταν, ήρθε, όταν είχαμε αυτή την ιδέα για αυτή την έκθεση, ίσως το πλαίσιο ήταν διαφορετικό. Το πλαίσιο τώρα έχει αλλάξει. Για καλό και ακόμα δεν ξέρω. Όμως η Κομισιό αυτή τη στιγμή θέλει να έχει μία στρατηγική. Επομένως, η έκθεση σας θα είναι η έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Άρα πρέπει να αναφέρεται σε όλα τα θέματα. Όχι λεπτομερώς, αλλά θα πρέπει να προσανατολίσει την, ε, την Επιτροπή για το ποια θα είναι η κατεύθυνση της στρατηγικής. Και αν το μέγεθος της έκθεσης ε, αποτελεί ένα πρόβλημα, γιατί το άκουσα ότι υπάρχει ένα τέτοιο πρόβλημα, θα πρέπει να ζητήσουμε την άδεια. Να, να παρεκκλίνουμε, αν θέλετε, από τις ε, για το μέγεθος, από τις διατάξεις για το μέγεθος. Διότι μιλάμε για μια στρατηγική που αφορά τους Ρωμά τα επόμενα χρόνια και αυτό θα πρέπει να το αναφέρετε και εσείς ε, στην μελέτη σας. Αυτό που αναφέρετε τώρα για την συλλογή ε, δεδομένων ε, και στοιχείων, τι, είναι, τι εννοείτε, θέλετε στοιχεία για το πόσοι είναι οι Ρωμά. Ευχαριστώ η Άννα Γκόμες. Ευχαριστώ και εκτιμώ ιδιαίτερα την μελέτη σας. Εγώ είμαι από την Πορτογαλία, δεν συμπεριλαμβανόμαστε στην έκθεση, στη μελέτη αυτή, συγγνώμη, αλλά επειδή υπάρχουν κάποιες εμπειρίες, και όσον αφορά την πολιτική θέληση εφαρμογής των πολιτικών, ε, ναι, όντως χρειαζόμαστε μια ευρωπαϊκή στρατηγική. Αλλά δεν αρκεί αυτή η στρατηγική, η κοινωτική στρατηγική. Χρειάζεται και πολιτική θέληση σε εθνικό επίπεδο για να εφαρμοστεί αυτή η κοινωτική ε, στρατηγική. Εγώ δεν είμαι ε, Ισπανίδα, εγώ είμαι Πορτογαλίδα, αλλά μπορώ να πω ότι στην Ισπανία είχαμε αυτή την επιτυχία, διότι οι Ισπανοί είχαν την πολιτική θέληση να εφαρμόσουν κάποια πολιτική. Λοιπόν, καλό είναι να έχουμε μια κοινοτική στρατηγική, αλλά πρέπει να έχουμε και σε εθνικό επίπεδο τα συγκεκριμένα εργαλεία. Εμείς ε, ε, στη χώρα μου δουλεύουμε πάρα πολύ καλά με τους διαμεσολαβητές που τους χρησιμοποιούν με τα κοινωτικά χρήματα. Σε έναν τομέα όμως που δεν, όπου επικρατεί μια κάποια σύγχυση και θα ήθελα να ακούσω την άποψη των επιρογνωμόνων είναι η εκπαίδευση για τα θέματα φιλετικών διακρίσεων, διακρίσεων ανάμεσα δύο φύλλα μάλλον. Υπάρχει μια σύγχυση στη χώρα μου. Δηλαδή, θα πρέπει να έχουμε σχολεία που θα θα, υπάρχουν, θα πηγαίνουν παιδιά τα οποία ναι μεν είναι ενταγμένα στην υπόλοιπη κοινότητα με τα παιδιά αλλά που θα πρέπει να είναι ε, σύμφωνα με, τους, ε, με, τις, ε, με αυτά που ζητάνε οι Ρωμά είναι, να, είναι ξεχωριστά αρένουν και θηλαίων τα σχολεία. Αυτό είναι αντίθετο με τη δική μας νομοθεσία, όμως οι Ρωμά για να πάνε τα κορίτσια στο σχολείο θέλουν να είναι θηλαίων. Άρα μήπως να κάνουμε μια υποχώρηση για να πηγαίνουν και τα κορίτσια στο σχολείο. Ευχαριστούμε. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω να ευχαριστήσω για την μελέτη αυτή που μας παρουσιάσατε. Είναι πολύ πλούσια σε στοιχεία. Κοιτάξτε, η κοινωνική και οικονομική πτυχή είναι παρούσα στη Ρουμανία. Δεν μπορούμε να ιεραρχήσουμε αυτές τις δύο διαστάσεις του προβλήματος, αλλά εγώ θα αναφερθώ σε μια άλλη πτυχή που έχει να κάνει με την χώρα μου, τη Ρουμανία. Όπως έλεγε και η συνάδελφος Άννα Γκόμες, υπάρχει η πολιτική βούληση σε όλα τα επίπεδα. Και σε κεντρικό επίπεδο και στα περιφερειακά και στα τοπικά επίπεδα. Και αυτό μπορεί να μπορούν να το επιβεβαιώσουν όλοι οι ευρωβουλευτές που πήγανε στην Ρουμανία για να δούνε την κατάσταση εκεί. Όμως υπάρχει και άλλο πρόβλημα στη Ρουμανία. Πώς μπορούμε να έχουμε ειδική στρατηγική για τους Ρώμα, ξέροντας ότι οι περισσότεροι άνθρωποι στη χώρα είναι φτωχοί εξαιτίας της γενικότερης οικονομικής κρίσης. Πώς να έχουμε ειδικά σχολεία στη Ρουμανία όταν τα παιδιά των Ρουμάνων εγκαταλείπουν το σχολείο. Πώς να μιλήσουμε για ειδικέ θέσεις απασχόλησης για τους Ρώμα όταν δεν υπάρχει απασχόληση στη Ρουμανία. Η κατάσταση υγείας επίσης πηγαίνει πολύ άσχημα στη Ρουμανία, όπως επίσης και το θέμα της στέγασης. Συνεπώς, μια τέτοια στρατηγική πρέπει να συνδέεται άμεσα με τη στρατηγική 2020 που μιλάει για τη μείωση της ανεργίας και για την ε, μείωση της εγκατάλειψης πρόωρα του σχολείου. Στη στρατηγική μας επίσης πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη σημασία σε κάποιες χώρες και σε κάποιες περιφέρειες της Ευρώπης που είναι ιδιαίτερα ευάλωτες οικονομικά. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Κορνέλη Εστ και μετά η Σεσίλια Βιλκστρόμ. Ευχαριστώ για την μελέτη αυτή. Πιστεύω ότι μας ε, έχει κάποια προοδευτικά στοιχεία. Θα αναφερθώ σε τρία σημεία. Καταρχάς, στη νομοθετική βάση θα ήθελα να σκεφτούμε ενδελεχώς ένα θέμα βασικό. Πρέπει να αλλάξει η νομοθεσία, το νομοθετικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ορισμένα θέματα ή όχι. Δεύτερον, χρειαζόμαστε ένα συγκεκριμένο δίκαιο για τους Ρώμα, ειδικά για τους Ρώμα ή όχι. Ή θα πρέπει εθνικά δίκαια να προσαρμοστούν σε συγκεκριμένε ανάγκες των Ρώμα. Θα ήθελα λοιπόν να ξέρω από εσά. Πρέπει το κοινοτικό δίκαιο απαιτεί, απαιτεί ορισμένες προσαρμογίες ή αυτό θα πρέπει να γίνει ε, στα, στα δίκαια και στις νομοθεσίες των κρατών μελών, στις συγκεκριμένε χώρες δηλαδή που έχουν Ρώμα. Πιστεύω επίσης ότι χρειαζόμαστε μια ζητή πολιτική, δηλαδή ενσωμάτωση και όχι διαχωρισμό στο Ρωμά, ε, ιδίως στα σχολεία. Στα σχολεία θα πρέπει να φροντίσουμε για την ενσωμάτωσή τους και όχι να ε, ξεκινήσουν ξεχωριστές ε, τάξεις για τα παιδιά το Ρώμα. Απ' την άλλη πλευρά όμως, στην παιδεία θα πρέπει να γίνουν ορισμένες αλλαγές ε, που, είναι ευρύτερε. Δηλαδή, στο μάθημα της ιστορίας, παραδείγματο χάρη, θα πρέπει να ενσωματωθεί η ιστορία των Ρώμα ή να γίνουν απαραίτητες αλλαγέ σε περίπτωση που υπάρχουν ασάφειες ή, ή λανθασμένες Πρέπει λοιπόν να ασχοληθούμε οπωσδήποτε με το θέμα της, ε, των διακρίσεων. Ορισμένες ε, ε, ομάδες Ρωμά υποφέρουν τόσο πολύ επειδή η επίσημη, το επίσημο κράτος υποστηρίζει διακρίσεις είτε στη σχολική εκπαίδευση είτε στην νομοθεσία. Γι' αυτό ε, πιστεύω ότι λείπει ο πέμπτος πυλώνας από τους τέσσερις που αναφέρεται, λείπει ο πυλώνας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αυτό πρέπει οπωσδήποτε να το συμπεριλάβετε. Και τέλος πιστεύω ακράδαντα ότι τίποτα δεν θα επιτύχουμε και τίποτα δεν θα γίνει εάν δεν επιτύχουμε την συμμετοχή των Ρώμα από το πρώτο βήμα. Εάν στην διαμόρφωση της στρατηγικής δεν συμμετάσχουν και οι θυγόμενοι δεν θα επιτύχουμε τίποτα. Δεν είναι δυνατόν να είναι εκτός ε, στρατηγικής. Γι' αυτό τα άτομα και οι σύνοντες οι οποίοι διατυπώνουν και διαμορφώνουν τη στρατηγική πρέπει οπωσδήποτε να συνεργαστούν μαζί τους. Ευχαριστώ πάρα πολύ η Σεσίλια Βίκστρομ καταρχάς και παρακαλώ ένα λεπτό θα σας δώσω για να σεβαστούμε το χρόνο μας. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Δεν υπάρχουν σουηδικά, δεν υπάρχει διερμηνία. Δεν έχουμε μετάφραση από σουηδικά. Εντάξει, θα συνεχίσω αγγλικά τότε, λέει η κυρία Βίλστον. Σας ευχαριστώ, ωραία. Λοιπόν, θα, θα μιλήσω αγγλικά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που παρουσιάσετε αυτή την έκθεση. Όπως είπε και η συνάδελφός μου, η έκθεση αυτή τονίζει ε, τα κοινωνικο-οικονομικά στοιχεία. Όμως πρέπει επίσης να ε, προβάλλουμε την ιστορική πτυχή, διότι η ιστορία μας διδάσκει πώς καταλήξαμε στην παρούσα κατάσταση. Έτσι μαθαίνουμε μέσα ιστορικών γεγονότων. Και αν γνωρίζουμε το ιστορικό υπόβαθρο, μπορούμε να ε, διαμορφώσουμε και το μέλλον. Στη χώρα μου, στη Σουηδία, πολλοί ζητούν μια, ε, τη δημιουργία μιας επιτροπής αλήθειας, δηλαδή πώς έχουμε εμείς αντιμετωπίσει και μεταχειριστεί τους Ρώμα από το 17ο αιώνα. Από τότε η μειονότητα αυτή έχει υποστεί διακρίσεις και αυτές οι διακρίσεις δεν έχουν ποτέ σταματήσει. Γι' αυτό πιστεύω ότι η ιστορική πτυχή είναι απαραίτητη και σας ενθαρρύνω να την εσωματώσετε στην έκθεσή σας. Το ψήφισμα το οποίο εμείς έχουμε υποβάλει στην αρχή του χρόνου στην, ως κοινοβούλιο ε, είναι σημαντικό και θα ήθελα να ρωτήσω την εισηγήτρια αν έχετε διαβουλευτεί με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για το θέμα των Ρώμα. Ορισμένες φορές τα μέτρα τα οποία λαμβάνουμε είναι σαν ένα... Ε, είναι συντόνιστα, δηλαδή παίρνουμε από εδώ και από εκεί διάφορα μέτρα και τα κολλάμε σε ένα, μέσα σε ένα πλαίσιο. Αλλά πρέπει εμείς να προετοιμάσουμε μία συγκεκριμένη οδό, έναν μονόδρομο δηλαδή πολιτικής και όχι διάφορες τεμαχισμένες πολιτικές. Η κυρία Αλφάνο. Δεν θα ήθελα να επαναλάβω ε, αυτά τα οποία είπαν οι προλαλήσοντες που με κάλυψαν στις παρατηρήσεις μου, φαίνε, μου φαίνεται ότι η έκθεση αυτή περισσότερο οικονομική. Έχει δηλαδή δώσει το βάρος ε, σε οικονομικά θέματα. Ε, Δηλαδή κάπως δίνει την εντύπωση ότι η ασωμάτωση των Ρώμα είναι σημαντική διότι θα βοηθήσει την ευρωπαϊκή οικονομία. Δεν νομίζω ότι αυτό είναι ο στόχος της ε, συνθήκης για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Εγώ θα περίμενα περισσότερο, να ακούσω περισσότερο για τη νομική βάση της αντιμετώπισης των Ρώμα, για τα στοιχεία, δεδομένα δηλαδή, ε, Παραδείγματο χάρη 8.600 Ρώμα που εκδιώχθηκαν, απελάθηκαν από τη Γαλλία προς τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία. Στοιχεία δεδομένα θα ήθελα να ακούσω. Ε, αυτό το στοιχείο το έχουμε και είναι ένα γεγονό που συνέβη από την αρχή του χρόνου. Επίση τι γίνεται στην Ιταλία. Ε, στην Ιταλία χτες δεν οι αρχές ε, στο Μιλάνο αρνήθηκαν την παροχή ε, εργατικών κατοικιών ε, στο Ρώμα και δεν τους έδωσαν καμία δυνατότητα προσφυγής κατά της απόφασης αυτής. Αυτά είναι θέματα νομικά τα οποία μας απασχολούν και θα περίμενα να ακούσω περισσότερα για αυτά τα γεγονότα. Ίσως θα έπρεπε να ρωτήσω την εισηγήτρια θα επισκεφθείτε τα κράτη-μέλη αυτά, την Γαλλία, την Ιταλία, τη Ρουμανία, να διαπιστώσετε επί τόπου τι συμβαίνει. Θα ζητήσετε από τα κράτη-μέλη να επιβεβαιώσουν αυτά τα στοιχεία. Και τέλος, κύριε Πρόεδρε, το ρωτώ αυτό γιατί σήμερα το πρωί μαζί με άλλους συναδέλφους ήμουνα στην συνεδρίαση που και διαπίστωσα την έντονη πολιτική βούληση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να διαπραγματευτεί ε, συμφωνίες ε, με χώρες όπως η Λιβύη. Ήμουνα στη συνεδρία στη Μαγκρέπ το πρωί και είδα ας πόσο έντονη είναι επισημία σύναψη συμφωνίες με τη Λιβύη και ρωτώ γιατί πρέπει να πάντοτε να προσέχουμε τόσο πολύ τις εξωτερικές συμφωνίες αφού, δεν μπορούμε να λύσουμε τα ε, ενίκο later on. There is one more contribution from uh, the side, and then we will ask you to uh, answer it. Uh, please, is the last. Τελευταία παρέμβαση από την κυρία Ματιά από του Ευρωβουλευτέ και μετά θα δώσουμε το λόγο πάλι στους προσκεκλημένου μα. Ευχαριστώ και ευχαριστώ και πάλι την εισηγήτρια. Όπως και οι συνάδελφοι πριν, έτσι και εγώ θέλω η μελέτη και η έκθεση αυτή να έχει τη θέση που της πρέπει. Ήρθε η ώρα να πάρουμε τα πράγματα στα χέρια μας. Και το Κοινοβούλιο, και το Συμβούλιο, και η Επιτροπή. Πολύ σύντομα, τρία στοιχεία. Πράγματι, ήρθε η στιγμή να εντάξουμε τους Ρώμα. Και τι σημαίνει να τους εντάξουμε. Σημαίνει ότι εμείς, σε επίπεδο κρατών μελών, πρέπει να φροντίσουμε για την ένταξη των Ρώμα, αλλά και εκείνοι από τη δική τους την πλευρά πρέπει να το θέλουν. Δηλαδή πρέπει εκατέρωθεν να γίνει ένα βήμα. Στην Ρουμανία προσπάθησα να καταλάβω την κατάσταση και πήγα επί τόπου. Και μου έκανε εντύπωση θετικά γιατί είδα ότι το κράτος, η Ρουμανία, κάνει ό,τι μπορεί για να ενταχθούν οι Ρώμα και σε επίπεδο εκπαίδευση και σε επίπεδο υγείας και φροντίζουν να υπάρχουν διαμεσολαβητέ και για τους δύο αυτούς τομείς. Όμως η Ρουμανία αντιμετωπίζει τεράστια προβλήματα που εμείς πρέπει να λύσουμε όσον αφορά την απορρόφηση των κοινοτικών κονδυλίων. Αυτό γίνεται όλο και πιο περίπλοκο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα έπρεπε να έχει ένα σύστημα διευκολύνσεων για τις νέες χώρες, Ρουμανία και Βουλγαρία. Θα μπορούσε η Επιτροπή να βοηθήσει αυτές τις χώρες να χρησιμοποιήσουν πιο εύκολα τα κοινωτικά κονδύλια. Βλέπετε, στη Ρουμανία υπάρχουν αν μη τι άλλο τρία μεγάλα προγράμματα για την ένταξη των Ρώμα. Είναι έτοιμα και τα τρία, αλλά μπλοκάρονται γιατί λείπουν μία-δύο υπογραφέ. Γι' αυτό προ Θεού η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ας φροντίσει να μην είναι τόσο περίπλοκα τα διαρθωτικά ταμεία. Τώρα, οι διαμεσολαβητέ που δουλεύουν στα διάφορα προγράμματα της Ρουμανίας βοηθούν πολύ. Το διαπίστωσα. Διαπίστωσα επίσης ότι οι μίξη στα σχολεία επίσης είναι κάτι που δουλεύει. Δεν είναι δυνατόν να έχουμε ένα σχολείο για Ρώμα και ένα άλλο για τους υπόλοιπους. Δεν ισχύει αυτό μόνο στη Ρουμανία. Πρέπει η Ρώμα, η κάνει, να αναμειγνύονται με τον υπόλοιπο ευρωπαϊκό πληθυσμό. Είτε πρόκειται για την υγεία, είτε πρόκειται για την εκπαίδευση. Καλά θα κάνουμε να φροντίσουμε να τους εντάξουμε, αλλά να φροντίσουμε και αυτοί να νιώσουν ελεύθεροι να ενταχθούν. Γιατί σίγουρα υπάρχουν πολλές αντιστάσεις και από τη δικιά τους την πλευρά. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Καλό θα ήταν να είχαμε περισσότερο χρόνο για να συνεχίσουμε, αλλά δεν έχουμε. Οπότε, δώστε μας τις απαντήσεις σας, παρακαλώ. Πατήστε το κουμπάκι και θα ανοίξει το μικροφόνο σας. Ευχαριστώ πολύ και την εισηγήτρια και τους ευρωβουλευτές εδώ για τα επικοδομητικά του σχόλια. Θα μας βοηθήσουν πάρα πολύ προκειμένου να συμπληρώσουμε την... Ναι, έχω πράγματι μερικά σχόλια, να που έχουμε λίγο χρόνο, θα είναι και λίγα και μετά θα δώσω το λόγο και στη συνάδελφο. Πρώτον, Λέτε ότι επικεντρωνόμαστε σε κοινωνικά και οικονομικά ζητήματα. Μα αυτό ζητήθηκε, αυτή ήταν η εντολή που είχαμε. Μας ζήτησαν να μην ασχοληθούμε με το θέμα της μετανάστευσης ή το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, διότι τα θέματα αυτά καλύπτονται σε άλλες εκθέσεις. Έτσι, λοιπόν, δεν μπήκαμε στα θέματα της μετανάστευσης και των διακρίσεων. Επίτηδες. Αυτό είναι ένα. Όντω, επικεντρωθήκαμε στα κοινωνικά και οικονομικά ζητήματα. Γιατί, Γιατί εμεί πιστεύουμε ότι εφόσον ενταχθούν στην ε, κοινωνική και οικονομική ζωή, βελτιώνεται το επίπεδο της ζωής τους και όπως είπε και κάποιος, αυτή είναι διαδικασία που παίρνει χρόνια, ίσως και 20 χρόνια. Συμφωνώ. Είπατε για τη Γερμανία χρειαζόμαστε καινούριου νόμους, πρέπει να σκεφτούμε σε άλλη βάση με ποιο τρόπο αντιμετωπίζουμε αυτά τα ζητήματα. Κατά τη γνώμη μου, ναι, έχουμε ένα μεγάλο και πολύ σοβαρό πρόβλημα που είναι το ότι εκατομμύρια άνθρωποι ζουν σε περιθώριο και σε συνθήκες που είναι απαράδεκτες σήμερα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα ναι, χρειάζεται μια διαφορετική προσέγγιση. Κάποιο μίλησε για σχέδιο Μάρσαλ. Ε, δεν ξέρω. Ίσως όπως το πρόγραμμα ΚΑΤΣ για την νοτιοανατολική ε, Ευρώπη μετά τον πόλεμο της Ιουγκοσλαβίας. Χρειάζεται δηλαδή μια μαζική παρέμβαση για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα των Ρώμα. Η συνάδελφος αναφέρθηκε πριν στη δυνατότητα δημιουργία μια Ευρωπαϊκή Υπηρεσία που θα ασχολείται ειδικά με τους τσιγκάνου με τους Ρώμα. Δεν έχουν χώρα, δεν τους εκπροσωπεί κάποια χώρα, οπότε η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να τους εκπροσωπεί. Μέσω, γιατί όχι, μιας ειδική υπηρεσίας η οποία θα ασχολείται με τα θέματα των Ρώμα. Και θα υποστηρίζεται βέβαια από την Ευρωπαϊκή Ένωση ολόκληρη για να εξυπηρετεί τους Ρώμα. Τέλος. Ότι η Ρουμανία είναι φτωχή χώρα. Ναι. Σίγουρα πολλά από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν ε, οι Ρώμα τα αντιμετωπίζουν και άλλοι Ρουμάνοι, οι Βούλγαροι πολίτες της χώρας τους. Σίγουρα δεν είναι θέμα προτεραιότητας. Το θέμα είναι ότι πρέπει και οι Ρώμα να έχουν την ίδια πρόσβαση στην Ρουμανία, στην υγεία, την εκπαίδευση, την απασχόληση, όπως και οι υπόλοιποι Ρουμάνοι πολίτες. Είναι πρόβλημα που συναντάμε σε πολλές ε, χώρες μέλη από τις χώρες που τελευταίες μπήκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έπειτα, το νομικό πλαίσιο. Ρωτήσατε. Κοιτάξτε, δεν έχουμε ειδικό τμήμα στην ε, μελέτη μας, προς το παρόν τουλάχιστον. Το στοιχείο κλειδί όμως εδώ είναι η οδηγία για την εφαρμογή της αρχής που μιλάει για ίση μεταχείριση ε, των ατόμων ανεξάρτητα από την ε, εθνη, εθνική τους καταγωγή. Είναι οδηγία του 2000. Σε αυτή τη βάση μιλάμε για μη διάκριση. Το πρόβλημα είναι όταν έχουμε να κάνουμε με κοινωνικές και οικονομικές πολιτικές ότι η κοινωνική πολιτική μετά τη Λισαβόνα εξακολουθεί να είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών. Αυτό είναι το ζήτημα. Και γι' αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο να έχουμε μια ευρωπαϊκή νομική βάση και γι' αυτό βασιζόμαστε μόνο στις διακρίσεις. Η συνάδελφός μου τώρα. Ευχαριστώ. Εν συντομία να προσθέσω κάποια σχόλια. Καταρχάς να ξεκινήσω από το ερώτημα που ετέθη για τη νομική βάση. Εμείς πιστεύουμε ότι πέρα του συγκεκριμένου στόχου αυτής της μελέτης, που είναι ευρύτερος ευρύτερος στόχος ε, και χρειαζόμαστε μεγαλύτερο ορίζοντα για να την αναπτύξουμε. θα πρέπει να δημιουργηθούν οι νομικές ε, δυνατότητες, να αναπτυχθούν οι στρατηγικές για τους Ρωμά, που και αυτό το επιτρέπει η συνθήκη της Λισαβόνας, ε, η οποία έχει διευρύνει την δυνατότητα να συζητήσουμε θέματα όπως η κοινωνική πολιτική παραδείγματος που έθιξε και ο συνάδελφος. Γιατί παραμένει εθνικό, εθνική αρμοδιότητα. Αυτό θεωρείται ένας κοινό τομέας ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη. Επομένως υπάρχει μεγάλο περιθώριο το οποίο μπορούμε να εκμεταλλευτούμε και το οποίο θα είναι χρήσιμο για να δημιουργήσουμε μια στρατηγική η οποία δεν ε, θα περάσει αναγκαστικά από, έναν δεσμευτικό, από μια δεσμευτική νομοθεσία, διότι η δεσμευτική νομοθεσία αφορά και απαιτεί απόλυτη πολιτική θέληση. Αυτό δεν να το ζητήσουμε τώρα. Είναι πολιτική, νομισματική, ανταγωνισμού και τέτοια. Εκείνο το, το, εκείνος εδώ μιλάμε για την στρατηγική που αφορά την περιθωριοποίηση, την φτώχεια κτλ. που δεν θίγουν μόνο τους Ρωμά αλλά και όλο ένα αυξανόμενο αριθμό ατόμων. Επομένως δεν μπορούμε να έχουμε ε, τέτοιου, τέτοιου είδους δεσμευτικές νομοθεσίες μόνο για τους Ρώμα. Χρειαζόμαστε κοινέ αρμοδιότητες Μοιρασμένε αρμοδιότητες ανάμεσα στα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στα κράτη. Ένα άλλο θέμα, το οποίο είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο, είναι η πολιτική θέληση που πολλοί έθιξαν. Χρειάζεται πολιτική θέληση από όλα τα κράτη-μέλη να δεσμευθούν να συγκεντρώσουν ε, τι στρατηγικές και τους πόρους για να εφαρμοστούν τα μέτρα αυτά. Και αυτό δεν μπορεί να γίνει από τη μια στιγμή στην άλλη. Υπάρχει δηλαδή επομένως η νομική βάση, αλλά χρειάζεται να, να βελτιώσουμε την θεσμική ικανότητα και τον συντονισμό. Αυτό χρειάζεται πολύ δουλειά. Κάτι άλλο για αυτά που ανέφεραν ε, οι συνάδελφοι, ε, διακριτική μεταχείριση, βασί θεμελιώδη δικαιώματα και παραδοσιακή αντιμετώπιση γενικότερα. Αυτό είναι αυτά είναι θέματα τα οποία δεν τα έθιξε η μελέτη, διότι δεν ήταν μέσα στις προδιαγραφές μας αν θέλετε. Όμως πιστεύουμε ότι θα πρέπει να γίνει δουλειά από όλου και από τα κράτη-μέλη και την Ευρωπαϊκή Ένωση, από τα θεσμικά όργανα δηλαδή, και άλλη δουλειά όμως πρέπει να γίνει από τους Ρωμά, τους ιδίους, από τους εκπροσώπους των Ρωμά, από τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις των Ρωμά, από τις πολιτικές οργανώσεις των Ρωμά, διότι η ιστορία, όλο το ιστορικό είναι ιδιαίτερα περίπλοκα και υπάρχουν ε, πολλοί παράγοντες που εμπλέκονται, κοινωνική, οικονομική, είχαμε, έχουμε διακριτικές μεταχειρήσεις, ε, ε, είμαστε λίγο μπερδεμένοι ανάμεσα στην, στο αίτιο και στο αιτιατό και από την φτώχεια περνάμε στις ε, διακρίσεις, στην περιθεριοποίηση, στην εγκληματικότητα, στην αντίδραση κτλ. Έχει δημιουργηθεί ένας φαύλος κύκλος και τον οποίο πρέπει να σπάσουμε και χρειαζόμαστε μια θετική αντίδραση όσον αφορά τις ε, θεσμικές ε, αρμοδιότητες που θα πρέπει να αναλάβουν και τα κράτη-μέλη και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν ιστορικές δυσκολίες, πολιτιστικές δυσκολίες, πολιτισμική ένταξη και εδώ για την ένταξη ε, είναι υπεύθυνη και τα, είναι και τα δύο μέλη. Οι, οι, κοινωνίες μας στην Ευρώπη είναι περίπλοκες, είναι προχωρημένες, οι κοινωνικοί κανόνες ε, είναι δύσκολοι και περίπλοκοι και για να είναι ειρηνική μας ε, η ζωή, για να γίνει η ειρηνική η ζωή μας πρέπει να τα δεχτούμε όλα αυτά. Και πρέπει να, σκεφ, να σκεφτούμε όλα αυτά και να τα δούμε. Ευχαριστώ. Λυπούμεθα απόλυτα. Λυπούμεθα πραγματικά γιατί δεν ε, είναι τόσο περίπλοκο το θέμα και που δεν μπορούμε να το εξαντλήσουμε. Πριν προχωρήσουμε στο επόμενο σημείο της ημερησίας διάταξης, θα ήθελα να ζητήσω από τον κύριο Μπάριστερ από την Κομισιό, μήπως θα ήθελα να πει λίγα λόγια. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Χωρίς μικρόφωνο κύριος Μπάριστερ. Λοιπόν, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους ε, για τη συνεισφορά τους. Ε, η Κομισιόν θα δημοσιεύσει την ανακοίνωσή της τον Απρίλιο του 2011 και πραγματικά περιμένουμε να συνεργαστούμε και με την ε, Προεδρία της Ουγγαρίας, όπως το κάναμε και με την Ισπανική Προεδρία και με τη Βελγική τώρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ τους κυρίους και την, τον κύριο και την κυρία από το LSE. Πραγματικά πιστεύω ότι η μελέτη τους είναι πάρα πολύ χρήσιμη, θα τη λάβουμε υπόψη μας και ευχαριστώ και πάρα πολύ τους βουλευτές, τους ευρωβουλευτές για όλες τις προτάσεις τους για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε πιο εύκολα και να χρησιμοποιήσουμε τα διάφορα ταμεία στα κράτη-μέλη κτλ. Πρόεδρος, ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ για την έκθεσή σας και τη συνδυσφορά σας, η οποία θα είναι πάρα πολύ χρήσιμη, ε, γιατί όπως βλέπετε έχουμε εργαστεί πολύ σκληρά για αυτή την έκθεση. Περνάμε τώρα στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης, που είναι η έκθεση για την κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και θα ήθελα να ζητήσω από τον εισηγητή Κίνγκα Γκάλα να κάνει, την εισηγήτρια συγγνώμη κυρία Γκάλα, να κάνει μια σύνοψη. Ευχαριστώ. Η πρώτη μας ανταλλαγή απόψεων έγινε τον Απρίλιο. Ένα λεπτό λέει η πρόεδρος να αποχωρήσουν όσοι θέλουν.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 Okay, I think we should we should start. Kinga, may I ask you to Ωραία, μπορούμε να συνεχίσουμε λοιπόν. Ε, συνεχίζει η συγγήτρια. Είχαμε την πρώτη ανταλλαγή απόψε, την πρώτη συζήτηση στο θέμα αυτό τον Απρίλιο. Και ήδη τότε Είχα, είχα σήξει θέματα τα οποία συνεχεία συζητήθηκαν δύο φορές με τον σκιώδη εισηγητή και τους συμβούλους των πολιτικών ομάδων. Σε, αυτή, σε αυτό το σχέδιο εξαίσεως έχω υιοθετήσει μία διαφορετική προσέγγιση και έχω εστιάσει στο θέμα από διαφορετικές οπτικές γωνίες. Το 2009 τέθηκε ενισχύ η συνθήκη της Λισαβόνας η οποία επέφερε σημαντικές βελτιώσεις στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ε, πιστεύω προσωπικά ότι μια τέτοια έξεση όπου κάνουμε μια αξιολόγηση των αλλαγών όπου αξιολογούμε τη νέα αρχιτεκτονική των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Πρέπει τώρα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να σκεφτεί, να μελετήσει αυτές τις αλλαγές. Μετά από τη συζήτηση με τους πολιτικούς συμβούλους και τους κοιόδης συζήτητες, συμφωνήσαμε να ακολουθήσουμε αυτή τη νέα προσέγγιση και να υιοθετήσουμε το νέο τίτλο και να συμπεριλάβουμε ένα κεφάλαιο για τις επιπτώσεις της συνθήκης της Λισαβόνας. Περιμέναμε βεβαίως και μια ανακοίνωση από την Κομισιόν. Η πως κυρία Ρέντιγκ, μου είχε υποσχεθεί ότι θα κάνει μια σχετική ανακοίνωση. Και επίσης είχα και την προθεσμία. Δυστυχώς έπρεπε να υποβάλω το σχέδιο εξέσεως πριν λάβω την ανακοίνωση, τώρα όμως έχω την ανακοίνωση της Κομισιόν, η οποία μπορώ να πω ακολουθεί βασικά την ίδια κατεύθυνση. Αλλά βεβαίως θα πρέπει να δεχθώ ορισμένε τροπολογίες οι οποίες αντανακλούν το περιεχόμενο αυτής της ανακοίνωσης. Το σημείο εκκίνησης ε, του σχεδίου εκθέσεώς μου αναφέρεται σε όλα τα προηγούμενα ψηφίσματα και τις συζητήσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, οι ερωτήσεις προς την Κομισιόν και όλα τα άλλα διαδικαστικά. Αλλά δεν αναφέρεται στο συγκεκριμένο περιεχόμενο κάθε άρθρου, αλλά αναφέρει μόνο τα σημαντικά. και βάσει του στόχου αυτής της έκθεσης αναφέρω κυρίως τις διάφορες εξελίξεις που έχουν σημειωθεί μετά την θέση ενισχύου της Λισαβόνας. Ε, στο ρόλο που θα παίξουν οι θεσμικές, ε, τα θεσμικά όργανα στη νέα αυτή αρχιτεκτονική για τα ανθρώπινα δικαιώματα και Αναφέρουμε επίσης στον ρόλο και στις εργασίες που επιτελούν άλλα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το πρώτο τμήμα της έκθεσης μου τονίζει τους τρεις πυλώνες του κοινοτικού συστήματος, του ευρωπαϊκού κοινοτικού, ε, του, του, συστήματος της Ένωσης, που είναι η συνθήκη της Λισαβόνας, δεσμευτικός χάρτης βεβαίως, και οι υποχρεώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τη Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και αναγνώριση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που αναφέρονται σε αυτή την σύμβαση. Και βεβαίως τρίτος πυλώνας είναι το κοινοτικό κεκτημένο το νομικό, νομοθετικό υπόβαθρο των κρατών μελών. Επίσης εξετάζω τους διάφορους φορείς, φορείς και τα ιδρύματα, τα όργανα τα οποία πρέπει να εφαρμόσουν αυτή την αρχιτεκτονική και αναφέρουμε στον τρόπο με τον οποίο εμείς ερμηνεύουμε το ρόλο της Κομισιόν τι καθήκοντα, τι εργασίες πρέπει να επιτελέσει η Κομισιόν, ποιος θα είναι ο ρόλος του Συμβουλίου, του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, του Κοινοβουλίου και των κρατών μελών. Αναφέρομαι δηλαδή στο ρόλο όλων των κοινοτικών θεσμικών οργάνων. Ε, σε ένα άλλο τμήμα του σχεδίου Εξέσεως αναφέρομαι στη συνεργασία με διεθνείς ε, οργανισμούς, με διεθνείς οργανώσεις, διότι και αυτό είναι σημείο κλειδί για να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε αυτήν την αρχιτεκτονική. Και αναφέρουμε επίσης ε, στην ε, βασική, στο βασικό ρόλο μας μέσα στο Συμβούλιο της ε, Ευρώπης και μέσα στον Οργανισμό Ενωμένων Εθνών. Στο τελευταίο μέρος της έκθεσης αναφέρουμε στις πιο σημαντικές προκλήσεις της νέας εποχής, διότι αυτό είναι ένα σημείο κλειδί. Εάν λοιπόν δημιουργηθεί ένα πλαίσιο θα πρέπει μέσα σε αυτό να ενταχθούν όλοι οι φορείς οι οποίοι καλύπτονται από τη νέα αυτή αρχιτεκτονική και οι οποίοι φορείς θα πρέπει να παίξουν το ρόλο τους ε, αντιμετωπίζοντας τις πιο πιεστικές προκλήσεις. Αυτές τις έχουμε αναφέρει αρκετές φορές στο παρελθόν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπό τη μορφή ψηφισμάτων ή μέσα στα πλαίσια συζητήσεων. Ε, αυτά εν συντομία έχω να πω για τη δομή του σχεδίου εξέσεως και μπορούμε να εμβαθύνουμε κατά τη συζήτηση και να μιλήσουμε ξεχωριστά για το ρόλο κάθε θεσμικού οργάνου, κάθε υπηρεσίας. Αυτό που θέλω να ξέρετε είναι ότι αυτή η έκθεση υπάρχει μόνο στα αγγλικά προς το παρόν, γαλλικά και αγγλικά και θα μεταφραστεί σύντομα σε όλες τις γλώσσες. Η προθεσμία υποβολής τροπολογιών είναι η 9η Νοεμβρίου και η ψηφοφορία θα γίνει. Το Νοέμβριο και ζητήσαμε μια έκτακτη συνεδρίαση της ομάδας για αυτό τον σκοπό. Γιατί αρχικά ο στόχος ήταν να ενταχθεί στην Ολομέλεια του Δεκεμβρίου, όπου θα μπορούσε να συχετιστεί με την ημέρα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Έτσι είχε προβλεφθεί αρχικά. Αυτές λοιπόν είναι οι τεχνικές διαδικασίες. Και όπως σας είπα στη συνάντηση με τους κοιόδους συγητές, θέλω να δω όλες τις τροπολογίες, ε, θα χαρώ ιδιαίτερα να τις μελετήσω και είμαι στη διάθεσή σας και πρόθυμη για κάθε συνεργασία για να καταλήξουμε σε ένα γενικά αποδεκτό κείμενο, αποδεκτό από όλη την Επιτροπή. Ευχαριστώ πολύ. Επαναλαμβάνει η πρόεδρος, 9 δεκάτου είναι η προθεσμία τροπολογιών και πρέπει, όπως και όλες οι άλλες εκθέσεις, να τη διαβάσετε και να υποβάλλετε τροπολογίες μέχρι την προθεσμία αυτή. Ε, η Μόνικα είναι πρώτη στο κατάλογο μιλητών. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ την συνάδελφό μου συγγήτρια που ανέλαβε και εσωμάτωσε όλες αυτές τις σημαντικές νομοθετικές αλλαγές στην έξεση της και συγχαίρω την κυρία Γκάλη ιδιαίτερα επειδή διευκρινίζει τον ρόλο των θεσμικών οργάνων ε, και πώς θα τον επιτελέσουν νέα αυτή η αρχιτεκτονική των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Δεν έχω ακόμα ε, υποβάλει τροπολογίες, θα ήθελα όμως να τονίσω ορισμένες πτυχές και να προτείνω ε, ορισμένα συμπληρωματικά στοιχεία. Δύο θέματα καταρχάς να τονίσω. Δύο θέματα τα οποία θεωρώ πολύ σημαντικά και που περιλαμβάνονται η συνθήκη της Λεσσαβόνας και η εποχή μετά την εφαρμογή δεν θα πρέπει μόνο να αντανακλά τα ανθρώπινα δικαιώματα και να ζητεί την εφαρμογή του, αλλά θα πρέπει να παίξει και πρωταρχικό ρόλο διεθνώς. διότι η συνθήκη αυτή είναι ένα θαυμάσιο νέο μέσον εφαρμογής ε, αυτών των δικαιωμάτων και της προώθησης της αποτελεσματικότητας και της εφαρμογής τους στα πλαίσια της εξωτερικής πολιτικής. Γι' αυτό πιστεύω ότι όλοι οι τομείς της εξωτερικής πολιτικής και διαθροτικοί τομείς θα πρέπει να, ενσωμα... να αναγκαλιστούν ε, ε, μια τέτοια ε, πολιτική ανθρωπίνων σε δικαιωμάτων. Δεύτερον, η έκθεση πολύ σωστά αναφέρει ότι μετά τη Λισαβόνα, Δημοκρατία και τα θεμελιώδη δικαιώματα έχουν προσλάβει μία νέα έκφραση στα πλαίσια της πρωτοβουλίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και έτσι η Ευρωπαϊκή Ένωση τώρα έχει τη δυνατότητα ανάλυσης πρωτοβουλειών για νέα, νέες νέες νομοθετικές προτάσεις. Και τέλος, ε, συμμερίζουμε τα συμπεράσματα της έκθεσης που ζητούν από τα θεσμικά όργανα να διπλασιάσουν τις προσπάθειές τους για την περαιτέρω ενημέρωση και συνειδητοποίηση των πολιτών έτσι ώστε να γνωρίζουν ακριβώς τα δικαιώματά τους και πώς να μπορούν να τα προασπίσουν. Επίσης, ε, θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε και να χρησιμοποιήσουμε την εμπειρία των δημοσίων οργανισμών και να εδραιώσουμε, να ενισχύσουμε τις σχέσεις μας με όλες τις συναφείς υπηρεσίες και τους συναφείς φορείς που ασχολούνται με αυτό το θέμα. Παρόλο που γενικά βρίσκω την έκθεση, το σχέδιο έκθεσης πάρα πολύ καλό και σωστό, θα ήθελα να προτείνω μερικές προσθήκες. Πρώτον, το θέμα της μετανάστευσης ιδίω ε, τα θέματα θεμελιωδών δικαιωμάτων των μεταναστών. Αυτό λείπει τελείω και το παρατηρητήριο δηλαδή λείπει τελείω από την έκθεση. Πιστεύω ότι η πολιτική μετανάστευση πρέπει να την, να, να την προσέξει περισσότερο η στην έκθεσή τη. Επίση δεν καλύπτεται από την έκθεση η, καταπολ... η, ο αγώνα, η μάχη κατά τη φτώχεια και του κοινωνικού αποκλεισμού. Αυτό και αυτό το θέμα λοιπόν στο σημείο του 95 θα ήθελα να αναφερθεί. Η δεύτερη προσθήκη αναφέρεται στο ρόλο ε, του Επιτρόπου που έχει τον τομέα των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων των πολιτών. Πιστεύω ότι ο Επίτροπος θα πρέπει τακτικά να προσκαλείται ε, στις συνεδριάσεις της Επιτροπής μας, της ΛΥΜΠΕ. Και ε, όμως πιστεύω ότι η διατύπωση του σημείου 14 θα πρέπει να διευρυνθεί διότι εκτός από τις διακριμένες δράσεις του Επιτρόπου η, το σχέδιο έκθεσης, θα πρέπει επίσης να αναφέρει το ρόλο του Επιτρόπου για τη βελτίωση της ενημέρωσης των πολιτών. Θα, για να μπορέσουν οι πολίτες να σεβαστούν τις ε, προσπάθειες που κάνει η Επιτροπή για την ε, δρέωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα πρέπει να οργανωθούν περισσότερες εκστρατείες ενημέρωσης έτσι ώστε οι πολίτες να ξέρουν πού μπορούν να προσφύγουν όταν θίγονται τα θεμελιώδη τους δικαιώματα. Ο Επιτροπής, παραδείγματο χάρη, θα πρέπει να εξηγήσει πότε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να παρέμβει και πότε δεν μπορεί να παρέμβει σε περιπτώσεις ε, παραβίασης ε, θεμελιωδών δικαιωμάτων. Δηλαδή, ποιες αρμοδιότητες έχει και ποιες δεν έχει. Μπορεί να παρέμβει μόνο μέσα στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα ήθελα επίσης να προτείνω μία αξιολόγηση ε, όλων των των νέων νομοθετικών ε, προτάσεων που έχουν, ε, άπτονται των θεμελιωδών δικαιωμάτων για να εξασφαλίσουμε ακριβώς ότι σέβονται το χάρτη δεν θα, πρέπει να εφαρμόσουμε μια πολιτική μηδενικής, ε, αντοχή, ε, μηδενικής ανοχής παραβίασης των διατάξεων του χάρτη ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ε, επιτροπή μια διαδικασία παρακολούθησης λοιπόν της σωστής νομοθετικής εφαρμογής ε, αυτές τις προτάσεις είχα να κάνω προσθήκη στην έκθεση και γενικά βρίσκω ότι η έκθεση αυτή είναι πάρα πολύ καλή και τέλος θα ήθελα να τονίσω ότι ναι, αυτή η αρχιτεκτονική θα αξιολογηθεί με το, ε, και κατά πόσο να εφαρμοστούν με το βάλιστο τρόπο τα θεμελιώδη δικαιώματα. Ευχαριστώ. Η κυρία Βέμπερ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για την δουλειά της. Ε, συναντηθήκαμε ε, ήδη αρκετές φορές η συγγήτρια και η Σκιώδης ε, και συμφωνήσαμε για το περιεχόμενο της έκθεσης που είναι μοναδική ούτως ή άλλως ε, και περιμένουμε από τη διάσκεψη των Προέδρων να εγκρίνουν την αλλαγή στον τίτλο και ελπίζω θα γίνει αυτό γιατί πιστεύω ότι ήρθε η στιγμή να εξετάσουμε τις αρμοδιότητες κάθε δομής της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά την θέση σε ισχύ της συνθήκης της Λισαβόνας. Αυτό θα βοηθήσει και το Κοινοβούλιο στις μελλοντικές του δραστηριότητες όταν αξιολογούμε την κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και όταν εξετάσουμε πόσο κάθε θεσμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, εκπληρεί τα καθήκοντά του. Η, βασιλή, βασική μου ανάγκη, αν θέλετε, είναι το Κοινοβούλιο, να, η βασική μου επιθυμία είναι να, συμφωνεί, να, παρα, να διατηρήσει το Κοινοβούλιο τις αρμοδιότητές του ε, και Θα υποβάλουμε βέβαια κάποιες τροπολογίες, αλλά οι περισσότερες από αυτές ε, αφορούν τα δικαιώματα αλλά και τις υποχρεώσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, αλλά το πόσο, πώς μπορούμε να προωθήσουμε και την δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα ε, και μέσω των σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις υπόλοιπες χώρες. Ίσως χρειάζονται και κάποιες γλωσσικές προσαρμογές για να είμαστε σίγουροι ότι δεν θα υπάρχουν παρερμηνίες ε, και τελικά το κείμενο να αποδειχθεί εις βάρος ε, όσων θέλουμε να υποστηρίξουμε. Λέγεται εδώ, ας πούμε, για, ε, θέλουμε να περιορίσουμε τις διακριτικές μεταχειρήσεις για ένα μεγάλο μέρος των μειονοτήτων. Αυτό μπορούμε να διαβάσουμε και από δύο πλευρές. Αλλά είναι, υπάρχει μια αμφισημία εδώ. Αλλά τέλος πάντων, σε γενικές γραμμές μπορούμε να πούμε ότι είναι καλή και συνεκτική έκθεση. Ευχαριστώ πολύ Ρενάτε. Ε, η Άννα Γκόμες, ε, η επόμενη μήτρια και η κυρία, και η, κυρία Σάρα Λάτφορντ είναι η επόμενη to uh, uh, report. Θα ήθελα να ευχαριστήσω ε, την Kinga ε, για την ε, έκθεση της πολύ καλή και είναι χρήσιμο σήμερα μετά την θέση σε ισχύ της συνθήκη της Χρυσαβόνας, να πούμε όλα όσα λέγονται στην έκθεση. Για να απαντήσω στο, στο έτοιμά σας να είμαστε σύντομοι, να διευκρινίσω για τρία θέματα. Θα δούμε αν θα γίνουν ε, τροπολογίες. Τέλος πάντων, θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να παρουσιάσουμε εδώ το όραμά μας. Δηλαδή ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι ένα σύνολο ε, ε, που αδιέρετο αν θέλετε, το οποίο όμως αποτελείται από κοινωνικά, οικονομικά και άλλα δικαιώματα. Και ίσως θα πρέπει να το διευκρινίσουμε ε, σε μια παράγραφο που δεν αναφέρονται π.χ. τα πολιτιστικά δικαιώματα. Επίσης στην παράγραφο 1 αναφέρεται στην παράνομη κράτηση των ε, μεταναστών. Αυτό αναφέρεται και στην παράγραφο 35. Δεν μπορούμε να αναφερθούμε στα ανθρώπινα δικαιώματα, στα θεμελιώδη και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ξεχνώντας ε, αυτά τα οποία έκανε η Ευρώπη ε, με την, ε, σε συνεργασία με τους Αμερικανούς για την ε, μεταφορά των κρατουμένων. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να υπάρχει στον κατάλογο και θα έπρεπε να αναφέρεται και στην παραγραφό 1 όταν μιλάμε για παράνομη κράτηση των ατόμων τέλο πάντων, εκεί θα πρέπει να μιλάμε και για βασανισμούς, διότι όντως βασανισμοί έγιναν. Επίσης στην παράγραφο 6 είναι καλή βάση εδώ που χρησιμοποιούμε, αλλά ίσως θα πρέπει να τονίσουμε ότι η πρόθεση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων συνδέεται και με την πρόθεση της δημοκρατίας. Αυτό πρέπει να το πούμε στην παράγραφο αυτή και να μιλήσουμε και για την εξωτερική δράση της κοινότητας. Και ίσως θα έπρεπε να διατυπώσουμε και την ανάγκη ότι η εξωτερική μας πολιτική δεν θα πρέπει να υποσκάπτει τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και σας παραπέμπω σε μια έκθεση του Human, Human Rights Watch που αναφέρεται στην Αιθιοπία. Η Αιθιοπία που παίρνει τη μεγαλύτερη βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση βοηθάει στην καταστολή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και όχι στην προώθηση και τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Επίσης, συμφωνώ απόλυτα μαζί σας για τον ρόλο του Κοινοβουλίου, ο οποίος θα πρέπει να ε, ενταθεί όσον αφορά την προβόθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Εμείς όμως έχουμε ζητήσει από την Lady Ashton να μας πει ε, ποια είναι η, συμφωνία, η εκείνη ώρα της συμφωνίας που διαπραγματεύθηκε με την Λιβύη και μέχρι στιγμή δεν μας έχει πει τίποτα. Και την επόμενη εβδομάδα θα βγει μια αντιπροσωπεία για τη Λιβύη. Και η συμφωνία μπαίνει στον στο τελευταίο στάδιο διαπραγματεύσεων. Επίσης στο σημείο 31 θα πρέπει να αναφερθούμε στις ε, συμβάσεις, στις συνθήκες. Η συνθήκη και η σύμβαση κατά των, ε, του, των βασανιστήριων είναι πάρα πολύ σημαντική. Επίσης συμφωνώ απόλυτα με αυτά που είπε η Μόνικα, ότι θα πρέπει να τα συνδέσουμε όλα αυτά και με την ε, μετανάστευση. Αυτά θα πρέπει να συμπεριληφθούν στο σημείο 35, στην παράγραφο 35. Θα πρέπει να αναφερθούμε και στις δράσεις ε, με την, ε, της, της συνεργασίας με την CIA. Τέλος πάντων όλα αυτά όσα έγιναν, τα σκοτεινά που έγιναν εκεί. Εκεί θα πρέπει να επαναθεωρηθούν όλες οι εξετάσεις still going on. And, uh, um, and finally, uh, I would... Παράδοσης τέλος πάντων ε, των ε, κρατουμένων και επίσης ε, οι συμφωνίες επανεισδοχής θα πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο διαπραγμάτευσης και αυτό συνδέεται επίσης και με την πολιτική ασύλου που θα πρέπει να εξεταστεί. Ευχαριστώ. Η Βαρόνη Λάντφορντ έχει τον λόγο και θα ήθελα να είστε σύντομοι γιατί δεν θα τελειώσουμε στην ώρα μας. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Φαίνεται ότι στην έκθεση έχουμε πολύ καλό υλικό. Ομολογώ ότι διάβασα πάρα πολύ γρήγορα και ούτε καν στα αγγλικά, στα γαλλικά. Um, I, I like, I like what's in it. Μου αρέσει αυτό που διάβασα και είναι σωστό που πρέπει να παρουσιάσουμε αυτή την σκηνή όπως έχει διαμορφωθεί μετά τη συνθήκη της Λισαβόνας ε, και θα πρέπει να δούμε ποιοι, ποιοι θεσμοί, ποια θεσμικά όργανα είναι υπεύθυνα για κάθε θέμα και στην παράγραφο 3 που αναφέρεται ότι η υπηρεσία θεμελιωδών ε, δικαιωμάτων αποτελεί τον εγγυητή για τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Ευρώπη. Αυτό δεν αποτελεί και εγγύηση, δυστυχώς. Στην παράγραφο 23 είναι αυτό και στην παράγραφο 3. Επίσης, αυτό που θέλω να πω είναι ότι τα τελευταία, όλα αυτά τα χρόνια που παρακολουθώ τις εργασίες της ε, Επιτροπής, ε, είχα κάποιες απορίες ε, για τις ε, εκθέσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, θεμελιδών δικαιωμάτων. Πιστεύω ότι θα πρέπει στην παράγραφο 35, αντί να αναφερθούμε στα διάφορα θέματα που αποτελούν ε, τις σύγχρονες προκλήσεις, θα πρέπει να αναφέρουμε έστω και ακροθυγός του τομείς που αντιμετωπίζουν ε, τα κράτη-μέλη δυσκολίες. Τίποτα όμως από όλα αυτά δεν γίνεται εδώ. Υπάρχει παράγραφος 1 που αναφέρεται στα θέματα που συζητάει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όμως δεν σχετίζεται αυτό με την παράγραφο 35 που αναφέρει απλώς και μόνο του τομείς όπου θα πρέπει να φροντίσουμε να παρακολουθούμε την πρόοδο. Δηλαδή στην έκθεση αυτή, εκτός του παράγραφου 1, δεν έχουμε κάποιες συγκεκριμένες ιδέες σχετικά με τους τομείς που δημιουργούν προβλήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και πιστεύω ότι κάπου θα πρέπει να ε, συμπεριλάβουμε και αυτούς τους τομείς που μας δημιουργούν αυτό το άγχος. Και συμφωνώ με αυτά που είπαν οι συνάδελφοι ότι θα πρέπει να αναφερθούμε στα θέματα ασύλου, επανεισδοχής, ε, επανυποδοχής, ε, παράδοσης και βασανιστήριων. Ε, επίσης θα λέμε ότι ή θα πρέπει να πούμε ότι είμαστε δυσαρεστημένοι γιατί ποτέ δεν μας είπαν τι έκαναν αυτές οι χώρες που συνεργάστηκαν στα προγράμματα αυτά. Το Συμβούλιο δεν μας απήντησε ποτέ. Επίσης, και βλέπω ότι η πρόεδρος μου κάνει νοήματα, τελευταία παρατήρηση, η διαφορά μεταξύ σοσιαλιστών, σοσιαλδημοκρατών και φιλελευθέρων. Οι φιλελεύθεροι πηγαίνουν στα κοινωνικά και δημοκρατικά, κοινωνικά και οικονομικά δικαιώματα, που όμως δεν μπορούμε να εκφράσουμε αριθμητικά το δικαίωμα στέγασης, ας πούμε. Τι σημαίνει αυτό. Τι σπίτι πρέπει να πάρεις. Δηλαδή, ε, δημιουργείς προβλήματα, γιατί τι σόι σπίτι ε, πρέπει να δικαιούσε, τι σόι δουλειά δικαιούσε. Δηλαδή, υπάρχει μια παράδοση, αν θέλετε, στη συγκεκριμένη περίπτωση ανάμεσα στους σοσιαλιστές και στους σοσιαλδημοκράτες. Ευχαριστούμε. Ο τελευταίος θα είναι ο κύριος Μπρόγκς ομιλητής και μετά θα κλείσουμε τη συζήτηση. Αλλά προηγουμένως από τους ε, πράσινους. Ευχαριστώ. Κοιτάξτε, πάντα έχω την ε, αίσθηση ότι κάτι λείπει. Εντάξει, το καταλαβαίνω. Πάντα λείπει κάτι. Και αντιλαμβάνομαι τις παρατηρήσεις. Όμως, εγώ θα σας μεταφέρω τέσσερις σκέψεις που είχε η ομάδα μας και που θα υποβάλουμε από μορφή τροπολογιών. Πρώτον, υπόθηκε, αλλά θέλουμε να επιμείνουμε περισσότερο στο πρώτο τμήμα. Θέλουμε να ανακουφίσουμε κάπως το ρόλο, όχι μόνο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αλλά και της Επιτροπής αυτής. Γιατί πολλές φορές, σε πολλές ευκαιρίες το έχουμε πει, αλλά πια έχει γίνει must. Πρέπει να το πούμε ότι εμείς ή ότι η Επιτροπή μας έχει να παίξει έναν βασικό ρόλο στα θεμελιώδη δικαιώματα. Και αυτό πρέπει να, είναι, να φαίνεται ρητά στο κείμενο. Είναι σημαντικό να γίνει μια σύνδεση ανάμεσα στις εσωτερικές πολιτικές και τις εξωτερικές επιπτώσεις της πολιτικής αυτής για τα θεμελιώδη δικαιώματα ή πώς η εσωτερική πολιτική επηρεάζει θεμελιώδη δικαιώματα. Δεύτερο τμήμα. Είναι σημαντικό να επενθυμίσουμε ότι οποιαδήποτε αξιολόγηση θεμελιωδών δικαιωμάτων πρέπει να συμπεριλαμβάνει και την Υπηρεσία Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, αλλά και συμπεράσματα από συζήτηση με την κοινωνία των πολιτών τέτοιες διαβουλεύσεις είναι πολύ βασικές. Πρέπει να υπάρχει συμμετοχή των μη κυβερνητικών οργανώσεων. Τρίτο, είναι η συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς. Πάντα είναι δύσκολο και το καταλαβαίνω. Έχουμε όμως καλά παραδείγματα συνεργασία με το Συμβούλιο της Ευρώπης, για παράδειγμα, για την εμπορία ανθρώπων και άλλα. τέλος, η παράγραφος 35. Αναφέρθηκε και πριν. Είναι καλή προσπάθεια, αλλά νομίζω ότι θα μπορούσαμε εδώ να προσέξουμε περισσότερο τις λίστες αυτές για το θέμα του πώς λογοδοτούμε. Αυτά τα πράγματα μπορούν να βελτιωθούν. Κατά τα άλλα, εντάξει, και εμεί είμαστε έτοιμοι να βοηθήσουμε και να είμαστε επικοδομητικοί στην παρετέρω συζήτηση. Ευχαριστούμε και τώρα τελευταία. Ο κύριος ε, Μπόξ έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Υπάρχουν αυτοί που υποστηρίζουν ε, τα δικαιώματα και αυτοί που όχι. Συνήθως κάθε κράτος θεωρεί ότι είναι δημοκρατικό. Τώρα, τα, οι ελευθερίες και τα κοινωνικά δικαιώματα που έχουν καθιδρυθεί στα κράτη τα τελευταία χρόνια δεν είναι κάτι που περιλαμβάνει, για παράδειγμα, την ελευθερία έκφρασης. Χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης κάνουν κηρύγματα υπέρ της δημοκρατίας, αλλά από την άλλη μεριά βάζουν στη φυλακή συχνά ανθρώπους που παραβιάζουν, μάλλον που, από τους οποίους θερούν την ελευθερία έκφρασης. Και αυτό δεν είναι θεωρητικό. Ο Γερτ Βίλτερς, για παράδειγμα, αυτή τη στιγμή διώκεται στην Ολλανδία. Γιατί? Επειδή εκαταδικάζει το δόγμα του Ισλάμ, όχι τους μουσουλμάνους. Αυτό θεωρείται απαράδεκτο. Τρεις χώρες έχουν διαπραγματευτεί και έχουν πάρει opt-out, όπως και το Ηνωμένο Βασίλειο, από τη Χάρτα Θεμελιωδών ε, Δικαιωμάτων. Παρ' όλα αυτά, διάφοροι υποστηρίζουν στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων ότι ίσως δεν υπάρχει αυτό το δικαίωμα, αλλά χωρίς να έχουμε καταλήξει σε κανένα συμπέρασμα. Βασιζόμαστε και σε έγγραφα του Συμβουλίου της Ευρώπης και σε αποφάσεις δικαστηρίων όπως του Λουξεμβούργου και του Στρασβούργου. Εγώ έχω ρωτήσει ξανά και ξανά. Αν υπάρχει μια διαφορά ανάμεσα στις αποφάσεις των δύο δικαστήριων για παράδειγμα, τι γίνεται, κανείς δεν ξέρει να μου απαντήσει. Ευχαριστούμε κυρία Κινκαλτόρη, συγγήτρια για τα σχόλιά της προκειμένου κλείσει η συζήτηση. Ευχαριστώ συνάδελφοι που ήσασταν επικοδομητικοί. Είπα ήδη στην εισαγωγή μου ότι είναι ευπρόσδεκτες οι τροπολογίες σας πρέπει να υποβάλλετε τροπολογίες για να βοηθήσετε να διαμορφωθεί καλύτερα η έκθεση αυτή. Οι περισσότερες από τις ανησυχίες σας είναι θεμητές, ορθές. Μπορούμε να τις συμπεριλάβουμε. Είναι καλές προτάσεις. Και βλέπω μάλιστα, κυρία Μπένοβα, για παράδειγμα, που θα μπουν οι δικές σας οι προτάσεις στο κείμενο. Το βλέπω ήδη. Υπογραμμίζω ότι η χάρτα θεμελιωδών δικαιωμάτων είναι δεσμευτική. Τα λέω αυτά στις παραγράφους 5 και 16. Πάντως ευχαριστώ πολύ για τις τροπολογίες. Κυρία Βίμπερ. Έχουμε ήδη συζητήσει μαζί. Αξίζει αυτή τη στιγμή να δούμε το θέμα των θεμελιωδών δικαιωμάτων από αυτό το πρίσμα. Βέβαια υπάρχει περιθώριο για τροπολογίες, το επαναλαμβάνω, Όμως υπάρχει εξήγηση, είναι διαφορετική εκδοχή αυτή που μιλάει για λιγότερες μειονότητες. Κύριε Γκόμες, συμφωνώ ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι αλληλένδετα. Στην παράγραφο 4 θα μπορούσε να περιληφθεί αυτό. Και φυσικά μπορεί να τροποποιηθεί και η παράγραφος 35. το να γίνεται μνήμα στις συμβάσεις είναι πάντα χρήσιμο, αλλά είναι επίσης πάντα δύσκολο να καλύπτουμε ένα μεγάλο εύρος θεμάτων. Πρέπει να δούμε ποιες είναι οι πιο σημαντικές συμβάσεις και να τις συμπεριλάβουμε. Για την κυρία Λάτφορντ. Για την υπηρεσία θεμελιωδών δικαιωμάτων. Δεν είναι εγγύηση. είναι θέμα παρατηρητηρίου ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αυτό ήθελα στο κείμενο. Η υπηρεσία μπορεί να προσφέρει στοιχεία στα θεσμικά όργανα που παίρνουν αποφάσεις. Γι' αυτό φτιάχτηκε η υπηρεσία αυτή. Όπως είπα και πριν, η παράγραφος 35 μπορεί να τροποποιηθεί. Κύριε Ρωμέβα, και εγώ σκέφτηκα να αλλάξω το ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εδώ. Αλλά ακριβώ επειδή ήταν μεγάλη έκθεση έπρεπε κάτι να κόψω και το κόψα. Αλλά ήθελα να το βάλω και θα προσπαθήσω και εγώ θα υποβάλω μια τροπολογία για να το επανεισάγουμε. Και οι διαβουλεύσεις με τις ε, με την κοινωνία των πολιτών. Είναι κάτι που θέλω και εγώ και συμφωνώ να βάλουμε την πλατφόρμα των μη κυβερνητικών οργανώσεων. Κύριε Μπρόντς, αναφερθήκατε σε κάποια θέματα. για τα οποία δεν μπορώ εγώ να σας απαντήσω για τους διάφορους μηχανισμούς. Πάντως, πολλά θέματα θα διευκρινιστούν και δεν θα αποτελούν εμπόδιο στην αρχιτεκτονική των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Σας ευχαριστώ πολύ όλους για την συνεργασία και ας συνεχίσουμε τη συνεργασία μας για να καταλήξουμε στις τροπολογίες. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, σε ευχαριστούμε πολύ Κίνγκα. Περνάμε στο επόμενο θέμα στην ενεμερήσια διάταξη που είναι η δημιουργία ενός δικτύου αξιωματικών συνδέσμων μετανάστευση. Συσυγητής είναι ο κύριος Τίας Δεμέρα. Ψηφίσαμε ενδεικτικά τον Απρίλιο. Έγινε άτυπος ο τριμερής διάλογος πριν από λίγες εβδομάδες. Πείτε μας λοιπόν παρακαλώ κύριε Συγητά, για την κατάσταση πραγμάτων Άντε, μισό λεπτό για να βγουν από την αίθουσα όσοι θέλουν να αποχωρήσουν. Okay, then, uh, Ωραία. Λοιπόν, κύριε Δίας Δεμέρα, σας ακούμε. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος. Όπως γνωρίζετε, η έκθεση αυτή έχει κρατήσει πάρα πολύ καιρό μέχρι να εγκριθεί. Έχουν γίνει μεγάλες συζητήσεις και με τις συζητήσεις αυτές έχουμε φτάσει στο τελευταίο στάδιο προκειμένου να εγκριθεί οριστικά η έκθεση αυτή. Χρειάστηκε πολύ γενναιοδορία από τους σκιώδεις συζητητές και από τους συντάκτες των τροπολογιών τους οποίους και ευχαριστώ πολύ. Όπως γνωρίζετε, πρόκειται για τροποποίηση του κανονισμού 377 του 2004 και συγκεκριμένα τα άρθρα 3, 4 και 6 του κανονισμού αυτού. Ξέρετε, η νομική βάση στην οποία βασιζόμαστε είναι το γράμμα Β του σημείου 3 των άρθρων 73 και 76 της Δεγματικής Συνθήκης της Ένωσης. Εδώ πρέπει να σας πω ότι όλοι γνωρίζετε πάρα πολύ καλά τι προβλέπει ο κανονισμός όσον αφορά τους υπαλλήλου. Ποιοι είναι οι στόχοι τώρα της τροποποίησης αυτής που θέλουμε. Είναι τέσσερις. Ο πρώτος μας στόχος είναι να αποφεληθούμε από τις αρμοδιότητες που έχουν οι αξιωματικοί αυτή σύνδεσης των 27 χωρών. Τα κράτη-μέλη έχουν αξιωματικούς συνδέσμους σε 133 χώρες στον κόσμο. Θέλουμε λοιπόν να μπορούμε να τους χρησιμοποιούμε με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο. Και θα σας πω πώς. Θέλουμε λοιπόν να αποφεληθούμε από τους αξιωματικούς ε, σύνδεσμους, να υποφεληθούμε από την πληροφορία και από την ανταλλαγή πληροφοριών μέσω του Econet και σας θυμίζω ότι το Econet, ανασφαλές ηλεκτρονικό δίκτυο πληροφοριών, δεν περιλαμβάνει ε, στοιχεία προσωπικού χαρακτήρα. Έπειτα θέλουμε ένα ταμείο για τα εξωτερικά σύνορα και θέλουμε επίσης και ένα σύστημα εξάμεινων εκθέσεων. Επαναλαμβάνω ότι ευχαριστώ από βάθος καρδίας την κυρία Γκυγιόμ, την Σιλβή πρώτα απ' όλα για τη συνεργασία της. Ευχαριστώ επίσης τον σταριμίρη Σέφε, την Φρανσίσκα Κέλλερ, τον ε, Ρουίθ Ταμπάρε, την Σεσίλια Βέλστρομ και την Ελέν Φλότρο, γιατί συνεργαστήκαμε στενά μαζί και με βοήθησαν να βελτιώσω το κείμενο. Όπως είπατε και εσείς κυρία Πρόεδρε, 13 Οκτωβρίου είχαμε έναν τριμερή διάλογο για να ενημερωθούμε για τη θέση του Συμβουλίου και της Επιτροπής όσον αφορά τις τροπολογίες που θα είχαν εγκριθεί εφόσον η ψηφοφορία που κάναμε δεν ήταν ενδεικτικού χαρακτήρα, αλλά πραγματική. Προτάθηκαν διάφορες τροποποίησεις με τέσσερις συμβιβαστικές τροπολογίες. Τις έχετε, στα αγγλικά τουλάχιστον φρόντισαν να σας μοιραστούν. Αυτές οι συμβαστικές τροπολογίες λοιπόν πιστεύω ότι καλύπτουν τις προσδοκίες, αν όχι όλων, αλλά τις περισσότερες που εξέφρασαν οι σκιώδες εισηγητές. Όπως γνωρίζετε, πρότεινα τέσσερις συμβαστικές και μία τροποποίηση στην αιτιολογική μου σκέψη. Αυτή η τελευταία, που είναι μεγάλη, έχει ως στόχο να καθορίσει με σαφή τρόπο και διαφυσβήτητο τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της, Ευρωπα... και της Επιτροπής Συνόμη Ελευθεριών του Πολίτη όσον αφορά την ορολογία που πρέπει να χρησιμοποιούμε όταν αναφερόμαστε στην λαθρομετανάστευση. Θέλουμε δηλαδή να φανεί η πρόθεσή μας. Να ξεχωρίσουμε τον όρο μετανάστευση από τον όρο λάθρο μετανάστευση. Διότι τέτοια διάκριση δεν υπάρχει στις ε, περισσότερες νομοθεσίες. Η πρότασή μου λοιπόν έχει να κάνει με τις τροπολογίες 1, 2, 4 και 6 και εν μέρη με την 8. Το κείμενο στο οποίο αναφέρομαι είναι ένα κείμενο το οποίο ετοιμάσαμε η Σιλβή και εγώ. Οι συμβαστικές τροπολογίες περιλαμβάνουν το πνεύμα και τις τροπολογίες 6 της κυρίας Γκυγιώμα και της 7 του κύριου Ταβάρες και των κυρίων Φλότρο και Κέλλερ, την 8 των κυρίων Φλότρο και Κέλλερ και τέλος περιλαμβάνουν και το πνεύμα της 9 της κυρίας Κέλλερ. Μετά από τις συζητήσεις που είχα με συναδέρφους από τους φιλελεύθερους, η τροπολογία 3 που αναφέρεται στην αλληλεγγύη μένει σε κρεμότητα. και επίσης οι πέντε της κυρίας Σκέλερ, όπου διαφωνεί το Συμβούλιο, διότι το Συμβούλιο πιστεύει ότι τα κράτη-μέλη δεν είναι υποχρεωμένα να ενημερώνουν το Κοινοβούλιο για θέματα που είναι δικιά του αποκλειστική αρμοδιότητας. Κατόπιν τούτων ζητάω από τους συναδέρφους να συμφωνήσουν με τις συμβαστικές τροπολογίες που έχουν στα χέρια τους, όπως επίσης και την τροποποίηση στην οποία αναφέρθηκα πριν, που έχει να κάνει με την οτιολογική σκέψη, έτσι ώστε να μπορέσουμε πια μια και έξω να εγκρίνουμε την έκθεση αυτή. Κύριε Πρόεδρε, σας παρακαλώ, δεδομένου ότι οι σοσιαλδημοκράτες έχουν δικαιολογημένες δυσκολίες για να ψηφίσουμε στις 15 του μηνός στην Επιτροπή μας προτείνω, ζητώντας τη γενοδορία όλων των πολιτικών ομάδων, να γίνει η ψηφοφορία ή δυνατόν μαζί με την έκθεση της κυρίας Κίνκαγκάλ στο Στρασβούργο τη Δευτέρα το βράδυ. Δεν λέω ότι πρέπει να αποτελέσει προηγούμενο, γιατί υπάρχουν άλλα προηγούμενα, το έχουμε ξανακάνει τόσες και τόσες φορές. Έτσι θα πετύχουμε τον στόχο της Βελγικής Προεδρίας, που συμμερίζομαι κι εγώ, να εγκριθεί η έκθεση αυτή στην Ολομέλεια του Δεκεμβρίου. Τίποτα άλλο. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ. Είναι αλήθεια ότι η ομάδα SMP θα έχει μία συνάντηση στη Βουδαπέστη και θα δούμε αν μπορεί να γίνει η ψηφοφορία έτσι όπως συζητήσαμε. Πριν προχωρήσουμε θα ήθελα να ε, ρωτήσω την κυρία Μπεν από την Προεδρία του Συμβουλίου αν θέλει να προσθέσει κάτι. Η κυρία Μπεν έχει το λόγο. Ευχαριστώ, λέει κυρία Δεμπρέιν. Πρώτα απ' όλα ευχαριστώ πολύ τον εισηγητή για τις συμβαστικές του τροπολογίες για την Προεδρία είναι το αποτέλεσμα επικοδομητικών συζητήσεων που είχαμε στον άτυπο τριμερή διάλογο στις 13 Οκτωβρίου. Βέβαια, δεν έχουμε συζητήσει με ολόκληρο το Συμβούλιο. Αυτές οι βαστικές ε, τροπολογίες είναι πολύ πρόσφατες, πρέπει να συζητηθούν ακόμα στο Συμβούλιο, αλλά πιστεύουμε ότι θα μπει το θέμα αυτό στην εμερήσια διάταξη της επόμενης ομάδας εργασίας που θα λάβει η χώρα στις 29 Οκτωβρίου. Οι συμβαστικές αυτές τροπολογίες πάντως πάνε σίγουρα προς τη σωστή κατεύθυνση όσον αφορά εμάς. Και πιστεύω επίσης ότι οι διάφορες αντιπροσωπείες θα συμφωνήσουν. Σας ευχαριστώ λοιπόν πολύ για τις συμβαστικές τροπολογίες κύριε Μέρα. Ελπίζω να εγκρεθούν εδώ και εύχομαι και εγώ, όπως και ο συγκητής, κάθε επιτυχία κατά τη διάρκεια της Βελγικής Προεδρίας ακόμα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα από την Ευρωπαϊκή Κομισιόν παρόντες είναι ο κύριος Νίλσεν και ο κύριος Ντόμπο, που θέλει να λάβει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και εγώ τον εισηγητή για την δουλειά του. Θέλω επίσης να εκφράσω τις ελπίδες μας για το ότι τα κράτη-μέλη στο Συμβούλιο θα δεχτούν τις συμβαστικές αυτές τροπολογίες και έτσι θα προχωρήσουμε. Ελπίζουμε επίσης η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να γίνει δεκτή όσο γίνεται πιο γρήγορα. Ωραία. Έχουμε τον κύριο Κέροπ και η Σεσίλια Ντίξον μετά, που θέλουν να συμμετάσχω στη συζήτηση. Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να συγχαρώ τον εισηγητή για την εργασία που έκανε και να καταστήσω σαφές ότι η υπηρεσία στήριξης ε, ασύλου, Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Στήριξη του Ασύλου. Είναι μια πάρα πολύ σοβαρή υπηρεσία που πρέπει να την βοηθήσουμε στι εργασίε της. Έχω μία επιφύλαξη μόνο. Πιστεύω σαφώς ότι προσπαθώντας να αντιμετωπίσουμε τέτοια ευαίσθητα ζητήματα πρέπει να μεγιστοποιήσουμε τη συνεργασία μας μεταξύ κυβερνήσεων και υπηρεσιών η νομοθεσία, νομοθετικές ρυθμίσεις και δομές δεν πιστεύω ότι αποδίδουν αυτά που πρέπει να αποδώσουν πάντοτε. Είμαι λίγο επιφυλακτικό. Αυτά, αυτές οι υπηρεσίες, αυτά τα γραφεία υπάρχουν και το κείμενο λέει ότι δημιουργείται ένα άτυπο δίκτυο. Είχαμε βεβαίως αξιωματούχους συνδέσμους μετανάστευσης και παλιότερα είχα μάλιστα ε, και εγώ επαφή με αξιωματούχους του δικτύου μετανάστευσης και αυτοί οι αξιωματικοί σύνδεσμοι ε, βοηθούσαν ε, στη συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς ε, όταν υπήρχαν αιτήσει παροχής ασύλου μετανάστευσης προς το Ηνωμένο Βασίλειο και ο ρόλος τους ήταν πάρα πολύ θετικός. Πιστεύω λοιπόν ότι αυτό το δίκτυο μπορεί να, είναι, να έχει θετικές επιπτώσεις εάν μπορέσουμε να ανταλλάξουμε απόψεις και εμπειρίες για τις βέλτιστες πρακτικές και εάν ε, μπορέσουμε αυτό το δίκτυο να το να επιτύχουμε να εργάζεται πιο αποτελεσματικά. Δεδομένου ότι το θέμα της ε, ε, της μη κανονικής μετανάστευσης ε, είναι της, είναι της μόδας. Ένας νέος όρος που χρησιμοποιείται τώρα στην Ευρώπη αντί της παράνομης μετανάστευσης. Αυτή η ερμηνεία, αυτός ο όρος δεν προσθέτει τίποτα το ιδιαίτερο πρέπει να είμαστε, ε, η αντικανονική μετανάστευση, πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί, πρέπει να προσέχουμε ιδιαίτερα ότι, διότι στόχος μας είναι όχι μόνο η ασφάλεια, αλλά θα πρέπει να φροντίσουμε και προς το συμφέρον των ετούντων ε, μετανάστευσης, ε, να διασφαλίσουμε τα δικαιώματά τους. Αλλά υπάρχουν και οι άλλοι οι οποίοι δεν τηρούν τις διαδικασίες, είναι παράνομοι και αυτό πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Και η χρήση ενός τέτοιου όρου, αντικανονική, αντικανονική μετανάστευση, αντικανονική διαδικασία, δημιουργεί περισσότερα προβλήματα παρότι επιλύει. Γι' αυτό έχω αυτή την επιφύλαξη. Εκτός τούτου, ο, ο, ο, ο έχει κάνει ένα εξαιρετικό έργο. η Ευχαριστώ. Το κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς πρέπει να πω ότι είμαι πλήρω αναπογοητευμένη που η μετάφραση στα σουηδικά δεν είναι διαθέσιμη. Παρακαλώ να καταγραφεί στα πρακτικά. Εν συνεχεία θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Ντίας Δεμερά για την εξαιρετική της εργασία και να τον ευχαριστήσω που συμπεριέλευε στο εξηγηματικό μνημόνιο τη δική μου τροπολογία. Εγώ θα ήθελα, ε, πρότεινα να αλλάξουμε το παράνομο σε αντικανονικό. Παράνομο ήταν σε αντικανονική. Δεν ήταν όπως δυνατόν να γίνει, δεδομένου ότι ο όρος illegal παράνομη ε, αναφέρεται στις συνθήκες. Όμως υπάρχουν περισσότερες πτυχές από την καθαρά, ε, καθαρή ερμηνεία του όρου παράνομη παρανομία σημειολογική ερμηνεία πρέπει να ληφθεί υπόψη, όπως επίσης και η νομιμότητα όταν χαρακτηρίζουμε ανθρώπους. Για μένα η πολιτική ερμηνεία είναι εξίσου σημαντική, δεδομένου ότι δεν θα δεχθώ ποτέ ότι ε, οποιοδήποτε άνθρωπος, οποιοδήποτε ανθρώπινο χαρακτηρίζεται παράνομο, δεν θα το δεχτώ αυτό ποτέ, και δεδομένου ότι με τον προλαλήσαντα μπορούμε να συμφωνήσουμε ότι διαφωνούμε, ε, προσβλέπω σε μια ενδιαφέρουσα συνεργασία με διαφορετικές απόψεις. Εδώ εμένω στην άποψή μου. Όταν οι τροπολογίες δεν μπόρεσαν να συμμετουθούν στην έκθεση, ο κύριος Δίας Τεμέρα ε, δέχτηκε στο επεξηγματικό μνημόνιο να, να αλλάξει τον όρο παράνομο σε αντικανονικό. Να καταβά δηλαδή μία προσπάθεια αλλαγής του, του όρου παράνομος ή παράνομη μετανάστευση σε αντικανονική και να προσπαθήσει αυτό να μπει ε, και στη συνθήκη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Σιγητά για την εργασία σας. Η Πρόεδρος, ε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα να ολοκληρώσω τον κατάλογο. Έχουμε τέσσερα μέλη. Παρακαλώ να είστε τηλεγραφική και επιτρέψτε μου να σας διακόψω, να σας κάνω ένα σήμα να, να ολοκληρώσετε δεδομένου ότι έχουμε και θα ήθελα λοιπόν, ήθελα να ευχαριστήσω καταρχάς και τον εισηγητή και ε, γιατί έλαβε υπόψη τις παρατηρήσεις των σκιωδών εισηγητών, όλε τις ανησυχίες μας, τις απόψεις μας. Ε, όντως έγιναν κάποιες τεχνικές αλλαγέ στο κείμενο. Ε, είναι περίπλοκο, οφείλω να ομολογήσω, και ενσωματώνει όμως μια καλύτερη ανταλλαγή απόψεων και με το Κοινοβούλιο και με το ΣΑΡ και με την ε, Υπηρεσία Μετανάστευσης ε, και πιστεύω ότι θα, δεν θα είναι τόσο ε, σκοτεινή όλη αυτή η συνεργασία, θα, είναι πιο, θα υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια. Διότι πραγματικά ε, εδώ με, την, ε, με το δίκτυο αξιωματικών συνδέσμων μετανάστευσης θίγονται και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Δεν μπορώ να ολοκληρώσω εδώ την ημέρα μας χωρίς να αναφερθώ και εγώ στο θέμα της ορολογίας το παράνομος αντικανονικός. Λυπάμαι γιατί δεν μπορέσαμε να ακολουθήσουμε όλο το δρόμο που, θα, θα ήθελα στο κείμενο που μας δώσαμε. Στο θέμα της παράνομης μετανάστευσης ε, εγώ πιστεύω ότι η διατύπωση αυτή δεν είναι σωστή. Η κυρία μου το ανέφερε και το θέμα της πολιτικής αξιολόγησης και εκτίμησης. Ε, ήθελα να πω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο για μένα να ακούω το επιχείρημα και μας το είπε το Συμβούλιο αυτό στον Τρίλογο ίσως ε, τα λέω πολύ γρήγορα, ε, ε, ότι το βασικό επιχείρημα που παρουσίασε το Συμβούλιο είναι «Μα έτσι το λέγαμε ανέκαθεν, άρα δεν μπορούμε να το αλλάξουμε». Αυτή είναι μια γραμμή την οποία εγώ δεν μπορώ να δεχτώ. Χαίρομαι που ο κύριος Ντεμέρα ευρήκε αυτή την, αυτό το συμβιβασμό, αν θέλετε, και πιστεύω ότι η ορολογία του σημειολογικά και πολιτικά είναι απόλυτα σωστή. Και είναι σίγουρο ότι θα υπάρξει συνέχεια σε αυτό το θέμα. Thank uh, Ευχαριστώ. Ο κύριος... Η κυρία Κέλλερ και μετά η Ρενάτε Βίμπερ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τον κύριο Ντίες Δεμέρα για τη θαυμάσια εργασία του στον τοσχέ αυτό. Δυστυχώς πρέπει να πω ότι θα αποσύρουμε τις ε, τροπολογίες μας ε, διότι δεν ε, συνάδουν με τους κανονισμούς και είναι πολύ κρίμα αυτό διότι είχαμε βασιστεί στην, στις διατάξεις του, των διεθνών οργανισμών και είναι ατυχές, ατυχής περίπτωση που ο κανονισμός δεν μπορεί να μας βοηθήσει σε αυτό Ίσως μπορέσει το Συμβούλιο στο μέλλον να λύσει αυτό το πρόβλημα, πάντως αποσύρουμε τις τροπολογίες μας. Όσον αφορά τώρα την ορολογία, και εγώ θα προτιμούσα λέμε αντικανονική και όχι παράνομη. Και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί το θέμα αυτό, διότι η προτίμησή μας είναι σαφής. Ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος, η κυρία Βέμπερ. Ευχαριστώ και εγώ θα ήθελα να συγχαρώ ε, τον κύριο Ντίας Ντεμέρα για την έκθεσή του. Αντιμετώπισε πολύ επικοδομητικά ε, τις ε, τροπολογίες και δέχτηκε αυτά που μπορούσε να δεχτεί, που είχε περιθώρια να δεχτεί. Όσον αφορά τώρα την ορολογία μεταξύ παράνομου και αντικανονικού, όταν συναντηθήκαμε στην Αμερική με τους Λατινοαμερικανούς φίλους μας, είδαμε πόσο δύσκολο είναι το θέμα αυτό εκεί, σε αυτό το μέρος του κόσμου. Υπάρχει νόμιμη, η νόμιμη πτυχή και η παράνομη πλευρά. Θα πρέπει λοιπόν να ενθετήσουμε μία επικοδομητική προσέγγιση, διότι εδώ το θέμα αυτό δεν αφορά μόνο την έκθεση, τη συγκεκριμένη, αλλά και πολλά άλλα θέματα. Δεν είναι οι άνθρωποι παράνομοι, είναι η κατάσταση μέσα στην οποία βρίσκονται παράνομοι. Θα μπορούσαμε ίσως με αυτή την παράφραση να ερμηνεύσουμε ότι με κανέναν τρόπο δεν εννοούμε ότι τα ανθρώπινα όντα, οι άνθρωποι αυτοί καθεαυτοί είναι παράνομοι, αλλά οι συνθήκες μέσα στις οποίες βρίσκονται. Ευχαριστώ, όλα η Πρόεδρος. Αυτή η συζήτηση ρολογίας ε, κανονικού, αντικανονικού, παράνομου και μη παράνομου ε, ε, δεν είναι μέσα στα πλαίσια τα σημερινά ήθελα και εγώ να κάνω μία παρόμοια παρατήρηση με τη Ρενάτα. Και στο παρελθόν αλλά και τώρα θεωρούσα ότι όταν λέμε παράνομη σε σχέση, χρησιμοποιούμε τον όρο παράνομοι με ανθρώπους, ε, ε, δεν είναι σωστό. Άλλο παράνομη μετανάστευση και άλλο παράνομοι μετανάστες παράνομη μετανάστευση είναι διαφορετική. Παράνομος μετανάστης εστιάζει στον άνθρωπο. Δεν είναι έγκλημα να περάσει κανείς ε, τα σύνορα παράνομα. Ε, είναι μία διοικητική παράβαση. Είναι μία ε, διοικητική παράβαση, αλλά δεν είναι ποινικό αδίκημα. Θα πρέπει λοιπόν να βρούμε ένα συμβιβασμό μεταξύ των όρων παράνομη μετανάστευση, αλλά όχι παράνομη μετανάστες. Ευχαριστώ. Ο κύριος ηγητής. Θέλετε να προσθέσετε κάτι. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα είμαι σύντομος. Όλα αυτά που συζητάμε έχουν να κάνουν με τον διάλογο με το Συμβούλιο. Θέλω να ευχαριστήσω το Συμβούλιο για τον ρόλο που έχει παίξει, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που ήταν τόσο γενναιόδορη και που είχε δραστήριο ρόλο. Κύριε Κύρχοφ, σας ευχαριστώ πολύ για τα λόγια σας. Πιστεύω ότι είναι πολύ καλό να βελτιώνουμε τις σχέσεις μεταξύ των κυβερνήσεων και των οργανισμών των υπηρεσιών. Τώρα για το θέμα αυτό του κανονικού ή αντικανονικού δεν συμφωνώ μαζί σας. <coughs> Και λυπάμαι που το λέω γιατί συμφωνούμε μαζί σε πολλά άλλα θέματα. Όμως εδώ θέλω να απαντήσω και στη Σεσίλια και στη Σιλβή και στην κυρία Κέλλερ, στη Ρενάτε και στη Σάρα Λάτφορτ. Εγώ δεν χρειάστηκε την αρχική μου θέση να την τροποποιήσω, γιατί η αρχική μου θέση, όπως όλοι γνωρίζετε, στην πολιτική μου ομάδα, αλλά και εκτός αυτής, είναι να χρησιμοποιώ πάντα τον όρο αντικανονικός και ποτέ παράνομος. Όπως ξέρετε, και αν δεν το ξέρετε σας το λέω να το μάθετε, η πιο πρόσφατη νομοθεσία σε θέματα μετανάστευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι στην Ισπανία του Νοεμβρίου του 2009. Στην ομοθεσία αυτή, με ένα περίεργο τρόπο, θα το πω έτσι, χρησιμοποιούνται και οι δύο όροι. Και όρος αντικανονική και όρος παράνομη μετανάστευση. Εμείς δεν τα πετύχαμε όλα, αλλά πετύχαμε να έχουμε μία συζήτηση σημασιολογική, νομική, αλλά και πολιτική για αυτό το θέμα. Και είπαμε ποια είναι η θέση μας, παρόλο που δεν το λέμε στην αιτιολογική σκέψη. Λοιπόν, κυρία Πρόεδρε, συμφωνώ για το ότι ο όρος δεν αφορά αποκλειστικά την έκθεση αυτή. Είναι μια ορολογία που αφορά και θα αφορά πολλές και διάφορες εκθέσεις και κείμενα. Αυτός όμως είναι ο δρόμος που πρέπει να ακολουθούμε κάθε φορά που κάπου εμφανίζεται σχετικός όρος, τώρα και στο μέλλον. Να το προσέχουμε και να προσέχουμε πάρα πολύ τι ορολογία χρησιμοποιεί τόσο το Κοινοβούλιο όσο και η Επιτροπή και το Συμβούλιο. Σας ευχαριστώ πολύ όλους. Ευχαριστούμε πολύ. Η συζήτηση ήταν πολύ ενδιαφέρουσα πράγματι. Πρέπει να συνεχίσουμε όμως τώρα με την ημερήσια διάταξη και το επόμενο θέμα που έχουμε είναι προ... πρόταση της Επιτροπής με εισηγητή τον κύριο Γιακολίνο για τις προποθέσεις εισόδου μόλις πικών τρίτων χωρών στο πλαίσιο επιχειρησιακής μετάθεσης. Έχετε το λόγο, παρακαλώ, από την Επιτροπή. Ε, Ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε το λόγο να σας παρουσιάσουμε την πρότασή μας. Η Επιτροπή πρότεινε κάτι όπως επίσης και για τους εποχιακούς εργαζόμενους. Στόχος μας είναι καλύτερη οργάνωση και πιο ελαστική πολιτική μετανάστευσης. Ελπίζουμε ότι με τον τρόπο αυτό θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε μια καλή μεταναστευτική πολιτική και ότι δεν θα είμαστε μόνο ένα οχυρό. Κατά τη γνώμη μας η πρόταση αυτή χρειαζόταν ήταν αναμενόμενη για να ενισχυθεί η οικονομία μας και να συμπληρωθεί με μέτρα που θα μας, που θα μας βοηθήσουν να πετύχουμε τους στόχους της στρατηγικής 2020. Οι ενδεπιχειρησιακές ε, μεταθέσεις αφορά άτομα υπηκός τρίτων χωρών. Είναι κάτι που έχει άμεση σχέση βέβαια με την μεταναστευτική μας πολιτική διότι μερικές φορές μας λείπει εργατικό δυναμικό ή θέλουμε να αντιμετωπίσουμε δημογραφικές δυσκολίες. Υπήκο λοιπόν τρίτων χωρών στα πλαίσιο της επιχειρησιακής μετάθεσης τα τελευταία χρόνια αποτελούν ε, έναν σημαντικό παράγοντα. Είναι προσωρινής διάρκεια οι μεταθέσεις αυτές και οι διαδικασίες που ακολουθούν οι πίκοοι τρίτων χωρών είναι διαφορετικές γιατί είναι διαφορετικοί μηχανισμοί που επικρατούν στα διάφορα κράτη-μέλη. Για να πάρουν άδεια εργασία, για παράδειγμα, οι διαδικασίες κρατάνε πάρα πολύ, είναι περίπλοκες. Και δυσκολεύονται τα άτομα αυτά να μετακινηθούν μεταξύ χωρών μελών. Και γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήρθε με την πρότασή της πρόταση η οποία αφορά υπηκόους τρίτων χωρών στο πλαίσιο επιχειρησιακής μετάθεσης. Πρόκειται είτε για καρτιζόμενους είτε για εργαζόμενους που πηγαίνουν από μια επιχείρηση στις χώρες τους σε μια επιχείρηση που ανήκει στον ίδιο επιχειρησιακό όμιλο αλλά βρίσκεται σε χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για τρία χρόνια το πολύ όταν πρόκειται για managers ή με ειδίκευση ή ένα χρόνο όταν πρόκειται για καταρτιζόμενους. Υπάρχουν ε, συγκεκριμένες ρυθμίσεις για τις οικογένειές τους για να διευκολύνεται επίσης η μετακίνηση των εργαζόμενων αυτών και μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα μέτρα που προτείνονται είναι εναρμόνιση των όρων ε, αποδοχής των ε, εργαζόμενων αυτών Μιλάμε επίσης για τη χρονική διάρκεια που πρέπει και αυτή να είναι εναρμονισμένη. Μιλάμε για την ε, πανένωση των οικογενειών, για την διευκόλυνση της κινητικότητάς τους μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τέλος θέλουμε και ένα συγκεκριμένο νομικό καθεστώς με άδεια διαμονής και εργασίας. Σύμφωνα με τη συνθήκη είναι τα κράτη-μέλη που έχουν την αρμοδιότητα για να αποφασίσουν ε, πόσα τέτοια άτομα μετατίθενται. Θέλουμε λοιπόν κοινού κανόνες και να μην υπάρχουν 27 διαφορετικά συστήματα. Οι επιχειρήσεις που βρίσκονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση έτσι μπορούν να καλύψουν καλύτερα και πιο εύκολα τις ανάγκες τους σε προσωπικό. Έτσι μπορούμε να πετύχουμε την οικονομία που θέλουμε τη βασισμένη στη γνώση και θα προσελκύσουμε και επενδύσεις ώστε να δημιουργηθούν περισσότερες θέσεις απασχόλησης στην Ευρώπη. Πιστεύουμε ότι η συζήτηση εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο θα καταλήξει σε μια ισορροπία και ελπίζουμε να έχουμε μια γρήγορη διαδικασία και το νέο αυτό μέσο μετανάστευσης να ταποκρίνεται στις ανάγκες των κρατών μελών και να προσφέρει και εγγυήσει ώστε να μην υπάρχουν καταχρήσεις. Ευχαριστούμε πολύ. Εκπρόσωπος της Βελγικής Προεδρίας τώρα. Παρακαλώ. Έχετε το λόγο, κύριε Άντερσον. Ευχαριστώ πολύ, Κυρία Πρόεδρε, θα είμαι σύντομη με αυτή την τόσο, μετά από αυτή την τόσο πλήρη παρουσίαση της Κομισιό. Αυτή η οδηγία ε, παρουσιάστηκε στο τελευταίο Συμβούλιο Τζάι και έγινε ευνοϊκά δεκτή από τα κράτη-μέλη που υπενθύμησαν και όπως ε, το έκανε και η Κομισιό, υπενθύμησαν την ανάγκη να προχωρήσουμε και στον τομέα της ε, νόμιμης μετανάστευσης. Η τεχνική εξέταση ξεκίνησε στην ε, Αρμόδια Επιτροπή τον Σεπτέμβριο όμως βρίσκεται ακόμα σε ένα πρώιμο στάδιο. Οι θέσει των κρατών μελών δεν έχουν καθοριστεί οριστικά. Οι περισσότερες αντιπροσωπείε ε, διατηρούν τι επιφυλάξει τους, επομένως είναι ιδιαίτερα πρόωρο αυτή τη στιγμή να καθορίσουμε την στάση του Συμβουλίου. Αυτό το οποίο σημείωσε η Προεδρία είναι το ότι το θέμα τη ενδοκοινοτική κινητικότητα ε, θέτει κάποια προβλήματα, γιατί πρέπει να τη δημιουργήσουμε καταρχά αλλά είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να συζητηθεί και αυτό θα γίνει στην επόμενη συνεδρίαση της ομάδας εργασίας. Η Βελγική Προεδρία έχει την πρόθεση να εργαστεί ε, σκληρά πάνω σε αυτό το θέμα και να ολοκληρώσει την πρώτη ανάγνωση έτσι ώστε να μπορέσουμε να εντοπίσουμε τις ε, βασικές δυσκολίες που υπάρχουν όμως λόγω του χρόνου που περνάει τόσο γρήγορα, ε, δεν νομίζω ότι η δική μας Προεδρία θα ολοκληρώσει την υιοθέτηση του φακέλου αυτού. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Η Ουγγρική Προεδρία θα το αναλάβει, θα αναλάβει τη σκητάλη. Κύριε Γιακολίνο, είστε ο εισηγητής μας. Ε, θα πάρετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε, άκουσα με ιδιαίτερη προσοχή και την παρουσίαση της Κομισιόν και της Προεδρίας. Προφανώς αυτή η πρόταση της οδηγίας εντάσσεται σε ένα πακέτο το οποίο αποτελείται από πέντε οδηγίες και που έχει σαν στόχο να ε, ρυθμίσει τα θέματα της ε, νόμιμης ενδοκινοτικής μετανάστευσης με την αγορά εργασίας. Ε, η οδηγία αυτή είναι πάρα πολύ σημαντική, διότι ε, οι ενδοεπιχειρησιακές μεταθέσεις ε, μπορεί να γίνουν και ανάμεσα στις τρίτες χώρες και στις κοινωτικές χώρες, αλλά μετά την πρώτη μετάθεση μπορεί αυτές οι κινήσεις να αφορούν τελείως την, αποκλειστικά το κοινοτικό έδαφος και αναφέρθηκαν σε αυτά τα θέματα και η Κομισιό όταν είπε ότι η διαδικασία με την οποία θα πρέπει να ρυθμιστεί η αίτηση αυτή είναι πάρα πολύ σύντομη. Έχουμε 30 μέρες περιθώριο και σε περίπτωση άρνησης θα υπάρχουν σημαντικά προβλήματα μετά. Ε, από το περιεχόμενο της οδηγίας αυτής ε, θίγονται πολλοί τομείς, παραδείγματος χάρη η επιστημονική έρευνα, διότι στο Κοινοβούλιο εξετάζεται η, η οργανική οδηγία που αφορά α, ε, τις επιστημονικές ανταλλαγές. Επίσης ε, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και, άλλα, και κάποια άλλα κριτήρια, όπως είναι η, οικογενειακή επανένωση. Επίσης θα πρέπει και εδώ να λάβουμε υπόψη μας ότι για θέματα επικουρικότητας προβλέπονται και κάποιες ε, ρυθμίσεις που θα μπορούσαν ε, να υιοθετήσουν τα κράτη-μέλη. Π.χ. ας πούμε τα κράτη-μέλη θα μπορούσαν να αποφασίσουν όσον αφορά την, την ροή των εργαζομένων. Τέλος πάντων υπάρχουν πολλές ε, δυνατότητες ε, και ούτως ή άλλως ε, δίδονται και δυνατότητες προσωπικής και επαγγελματικής ολοκλήρωσης, τρία χρόνια για τους μάνατζερ και ένα χρόνο για τους ειδικευμένους. Αυτές είναι προθεσμίες που θα πρέπει να τις ε, εξετάσουμε. Ε, στο Συμβούλιο ακούσαμε ότι υπάρχουν διαφορετικές απόψεις. Θα πρέπει να τις δούμε και αυτές και ίσως θα πρέπει να κάνουμε και κάποιες άλλες αξιολογήσεις, να επιτρέψουμε με κάποιες παρεκκλήσεις στην οικογενειακή επανένωση όσον αφορά τώρα τον ορισμό των ειδικών, των εξειδικευμένων θα πρέπει να το συζητήσουμε. Επίσης, ε, τον ορισμό του επιχειρηματικού ομίλου θα πρέπει να τον επανεξετάσουμε. Τέλος πάντων, επειδή και η αίθουσα είναι λίγο κενή, δεν χρειάζεται να πούμε και σε πολλές ε, λεπτομέρειες επί της ουσίας. Εδώ στον τίτλο αναφερόμαστε στις μεταθέσεις. Δεν, είναι, δεν, αφορά, δεν αφορά το κείμενο της μεταθέσεις αυτές καθεαυτές, διότι η μετάθεση σημαίνει ότι περνάει ε, κάποιος από μία επιχείρηση σε μία άλλη για όριστο χρονικό διάστημα. Όχι, εδώ μιλάμε για κάποιες αποσπάσεις που γίνονται για συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα. Τώρα, είμαι στη διάθεση όλων και των σκιωδών εισηγητών, εάν και εφόσον θα έχουν να κάνουν κάποια πρόταση, αλλά πιστεύω ότι το κείμενο αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό σε αφορά την, με τις μεταναστευτικές ροές και κυρίως τις μετακινήσεις των εξειδικευμένων εργαζομένων που πρέπει να γίνουν ε, σε σύντομο χρονικό διάστημα. Πρέπει να υπάρχει μια ταχύτητα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Υπάρχουν ε, κάποια μέλη που θα ήθελαν να κάνουν κάποιες παρατηρήσεις. Ε, η κυρία Χίρς πρώτα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πιστεύω ότι η οδηγία αυτή είναι ευπρόσδεκτη και ανταποκρίνεται ακριβώς και στα πρότυπα τα οποία χρειαζόμαστε στην Ευρώπη εν ώψη βεβαίως και των σύγχρονων μεθόδων εργασίας. Έχω μία ερώτηση. Η Κομισιόν ορίζει μία προθεσμία 30 ημερών. Από την άλλη πλευρά στην οδηγία έχουμε 90 μέρες για το αεροπορικό εισιτήριο. Θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω μήπως υπάρχει μία ασυμβατότητα μεταξύ των προθεσμιών 30 και 90 ημερών. Μήπως ε, θα πρέπει τα κράτη-μέλη να ξανασκεφτούν ότι οι αποφάσεις που λαμβάνονται εντός 30 ημερών να ανταποκρίνεται και στην πραγματικότητα είναι εφικτό δηλαδή να ληφθούν επιφάσεις σε 30 μέρες. Ευχαριστώ. Η κυρία, η Σεσίλια και μετά ίσως η κυρία Σμιτ να απαντήσει. Ευχαριστώ. Μιλώ εκ μέρους του συναδέλφου μου, του κυρίου Γιάν ο οποίος είναι άλλος και ηγητή που δεν μπόρεσε να είναι εδώ παρόν. Είμαστε ευτυχεί που βλέπουμε επιτέλους αυτή η τελική πρόταση της ε, Κομισιόν παρουσιάζεται στην Επιτροπή μας. Η πρόταση είναι πραγματικά σημαντική αν θέλουμε να ε, ολοκληρώσουμε μία ε, μεταναστευτική πολιτική και ο κύριος Γιάν Μόλτερς ε, ήθελε να τονίσει ότι δεν δίδουμε τις ε, ίδιες εγγυήσει ε, στους εποχιακούς εργαζόμενους. Δεν παρέχουμε λοιπόν το ίδιο πλαίσιο. Κατά τη δική του ερμηνεία δεν είναι βέβαιο αν καλύπτουν οι προτάσεις αυτές και τους εποχιακούς εργάτες και θα ήθελα να εκπονηθεί μια μελέτη σε αυτό το θέμα. Όσον αφορά τώρα τη διευκόλυνση των ενδοεπηρεσιακών μεταθέσεων, θα ήθελα να υποστηρίξω τον εισηγητή και να ευχηθώ εκ μέρους του κυρίου Μόλντερς και εμού μία ταχεία πρόοδο της εξέσεως. Πριν ολοκληρώσουμε, να ξαναδώσω το λόγο στην κυρία Σμιτ, άνετο το επιθυμεί. Ευχαριστώ. Όσον αφορά την μπλε κάρτα και την οδηγία για την μπλε κάρτα, οι ενδοεπιχειρησιακές μετασέσεις δεν καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή Μπλε Κάρτα. Εδώ πρόκειται για μια ταχεία διαδικασία σε περιορισμένο χρονικό διάστημα, διότι οι άνθρωποι αυτοί έρχονται μόνο για ένα πολύ περιορισμένο χρονικό διάστημα και γι' αυτό θέλουμε να δράσουμε μια διαδικασία η οποία να του επιτρέπει αυτή την ταχεία ε, ρύθμιση, την ταχεία περαίωση των διαδικαστικών ρυθμίσεων ευχαριστώ ιδιαίτερα όσους υποστήριξαν τις προτάσεις μας αυτές. Είμαι πολύ ευγνώμων. Η Πρόεδρος, ευχαριστώ. Θα προχωρήσουμε τώρα στο τελευταίο θέμα που έχουμε μία κοινή συζήτηση της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ευρωπαϊκής Ένωσης Ισλανδίας και Νορβηγίας σχετικά με την εφαρμογή ορισμένων διατάξεων της Σύμβασης ε, της 29ης Μαΐου 2000 και του προστατώμενου σε αυτή πρωτοκόλλου για την αμοιβαία δικαστική συνδρομή επιτονικών υποθέσεων μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα περιμένουμε μερικά λεπτά και Ο ένας, ο ένας είναι ο κύριος Μόραες και η άλλη είναι ο Ταβάρες. Είναι ο Ταβάρες. Ο Ρούι Ταβάρες, μάλιστα. Θα little Να περιμένουμε λίγο, λέει η Πρόεδρος. Ναι, ναι. Okay. Mr. Tavares, can, we start your report? you are here and then we can move. με κύριε Ταβάρες, μια εδώ, για να ξεκινήσουμε τη συζήτηση. και ο Ένα λεπτό. for some minutes? It's coming.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 Uh, από ό,τι μου λένε, ο εκπρόσωπος της Κομισιόν είναι εδώ. Θα συζητήσουμε και τις δύο εκθέσεις από κοινού. Θα ήθελα να σας ζητήσω ε, πρώτα να ζητήσω τον εκπρόσωπο της Κομισιόν να συνοψίσει τις απόψεις της Κομισιόν και μετά θα προχωρήσουμε στους συζητητές. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Όπως ξέρετε, εδώ ασχολούμεθα με δύο παλιές συμφωνίες που είχαν συναφή με την ε, Νορβηγία και την ε, Ισλανδία. Το, ε, μία αφορά την αμοιβαία δικαστική συνδρομή από το υποθέσεων μεταξύ των κρατών μελών τη Ευρωπαϊκή Ένωση στις 29η Μαου του 2000. Και το δεύτερο αφορά τη, μια γενικότερη διαδικασία παράδοση μεταξύ των κρατών μελών τη Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Ισλανδία και τη Νορβηγία. Είναι παλιέ συμφωνίε και υπογράφηκαν το 2003 και το 2004, δηλαδή αρκετό χρόνο πριν. Αλλά σύμφωνα με τα όσα ίσχυαν πριν από τη Συμφωνία της Συνταβόνα, τα κράτη-μέλη είχαν τη δυνατότητα να μπλοκάρουν τα, τα αποτελέσματα αυτής της έκθεση, αυτής της συνθήκης, τη συμφωνίας τέλος πάντων, ε, σύμφωνα με κάποιες εκκρεμότητες εσωτερικές, που θα μπορούσαν να πάρουν πολύ χρόνο. Λοιπόν, ε, κάποια κράτη-μέλη έκαναν την δήλωση αυτή το στο Συμβούλιο, γι' αυτό ακριβώς η, η, υιοθέτηση αυτής της συμφωνίας μπλοκ, μπλόκαρε για κάποια χρώματα. Εν τω μεταξύ όμως μπήκε σε εφαρμογή η συνθήκη της Ρεσαβόνας το 2009 και εδώ υπάρχουν νέοι κανόνες που εφαρμόζονται στα ε, αποτελέσματα των ε, διεθνών συμφωνιών ε, με τις ε, τρίτες χώρες. Και επίσης εμφανίστηκε ο καινούριο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Άρα όλες αυτές τις θέσεις είναι επιπαλαιωμένες. και όλα τα αιτήματα των κρατών μελών ότι θα έπρεπε δηλαδή τα κράτη-μέλη να ρυθμίσουν πρώτα τα εσωτερικά θεσμικά τους προβλήματα, όλα αυτά ακυρώθηκαν από το 2009. Γι' αυτό ακριβώς η Κομισιόν άμεσα θα έλεγα υπέβαλε μία πρόταση για, ένα, για μία απόφαση του Συμβουλίου σύμφωνα με τους νέους κανόνες ε, και ε, απαιτείται σύμφωνα με τους νέους κανόνες η έγκριση του Κοινοβουλίου. Και γι' αυτό θα συζητάμε εδώ, στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών Δικαιοσύνης και Ιστορικών Υποθέσεων, που θα πρέπει να γνωμοδοτήσει η Επιτροπή αυτή για να σας πω λίγα λόγια για το περιεχόμενο της, ε, των συμφωνιών αυτών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πολύ στενές ε, σχέσεις και συνεργασία και με την Ισλανδία και με την Νορβηγία, σε πολλούς τομείς. Και κυρίως στον τομέα της εσωτερικής αγοράς και του ανταγωνισμού. Επίσης, ε, τα κράτη αυτά ανήκουν συμφωνία Σέγγεν και, όπως θα δείτε, αμέσως το Σέγγεν, η ελεύθερη κυκλοφορία δίνουν την δυνατότητα στους πολίτες να κυκλοφορούν ελεύθερα στα εσωτερικά σύνορα της κοινότητας. Επομένως, οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει και που δημιουργεί αυτή, δημιουργούν αυτές οι συμφωνίες είναι οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν και τα κράτη-μέλη της ε, κοινότητας. Παραδείγματο χάρη τα θέματα εγκληματικότητας, που είναι ιδιαίτερα επίκαιρα. Επίσης, οι χώρες αυτές δεσμεύονται από τη Συμφωνία Σέγγεν και από ένα κομμάτι της Συμφωνίας Σέγγεν που ε, αφορά την αστυνομική συνεργασία. Τα περίφημα μέτρα αντιστάθμισης ε, τα οποία έχουν ε, συμπεριληφθεί στη Συμφωνία Σέγγεν. Όλα αυτά εξηγούν το λόγο για τον οποίο και οι δύο αυτές χώρες αλλά και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν ένα κοινό συμφέρον να ευθυγραμμίσουν ε, τις διατάξεις που αφορούν την αστυνομική συνεργασία και να υπάρχει μια πιο σύντομη και ευέλικτη ε, διαδικασία παράδοσης των ε, καταδίκων ή των ατόμων τα οποία αυτή τη στιγμή βρίσκονται ενώπιον των δικαστηρίων. Είπαμε ότι υπήρχε μια συμφωνία, μια συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορά την ε, Ισλανδία και την Νορβηγία λόγω ακριβώς της ε, συμφωνίας Σέγγεν. Όμως κάποιες άλλες διατάξεις δεν εφαρμόζονται και αυτό είναι ένα κενό το οποίο θέλουμε να καλύψουμε. Επομένω, παραδείγματο χάρη, σύμφωνα με την καινούργια συμφωνία του 2003, όταν και εφόσον ε, τεθεί σε εφαρμογή και ισχύσει, μετά από την έγκριση του Κοινοβουλίου και την απόφαση του Συμβουλίου και την ε, ανταλλαγή νομοθετικών ε, κειμένων, θα μπορούσε να υπάρχει συμφωνία ανάμεσα στην Ισλανδία και την Νορβηγία και οποιαδήποτε ε, αρχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, π.χ. για τους μάρτυρες κτλ. Αυτό το οποίο μπορούμε να κάνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούμε να το κάνουμε και με την Ισλανδία και την Νορβηγία. Τώρα, όσον αφορά την δεύτερη συμφωνία, η οποία είναι από το 2006, ακολουθεί το μοντέλο της Συμφωνίας για το Ευρωπαϊκό Ένταλμα, ακολουθεί δηλαδή τους μηχανισμούς ε, που ε, δημιουργούν το πλαίσιο για την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Εντάλματος, επιτρέπει την διαδικασία παράδοσης των, ε, των καταδίκων ή αυτών που δικάζονται. Η διαδικασία θα είναι πιο εύκολη υπάρχουν διατάξεις ε, που βασικά ε, αποτρέπουν οποιαδήποτε πολιτική παρέμβαση. Δεν υπάρχει, όπως ας πούμε για την έξινε στα θέματα έκδοσης και πολιτική ανάμιξη, είναι καθαρά απόφαση των δικαστηρίων. Βέβαια υπάρχει μια παρέκκληση από το, από το δεδικασμένο. Ε, και οι προθεσμίες που προβλέπονται είναι 10 μέρες ...αν υπάρχει σύμφωνη γνώμη του, του ενδιαφερομένου και 60 μέρες αν δεν υπάρχει. Ε, όλες αυτές είναι εξελίξεις ε, τις οποίες καλωσορίζει η Κομισιό. Αυτές οι συμφωνίες ε, αποτέλεσαν αντικείμενο διαπραγματεύσεων ε, πριν από πολλά χρόνια, άρα κάποια στιγμή πρέπει να, έρθει και ε, πρέπει να εφαρμοστούν και Χαιρόμαστε διότι η, συμφωνία της, η συνθήκη της Λισαβόνας θα δώσει ένα ενισχυμένο ρόλο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ενισχυμένο ρόλο για όλες τις διεθνείς ε, συμφωνίες. Σύμφωνα με το άρθρο 118 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα, εάν υπάρχουν ερωτήσεις, από το είμαι έτοιμος να απαντήσω και σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ. Thank you very much. Uh, before we move on... Ευχαριστούμε και συνεχίζουμε. Το Συμβούλιο τώρα. Θέλει το Συμβούλιο να μας πει κάτι γι' αυτό. Ναι. Πρώτα απ' όλα ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε το λόγο. Η Βελγική Προεδρία χαίρεται για την σύναψη αυτών των δύο συμφωνιών που είναι πολύ σημαντικές στα πλαίσια των σχέσεών μας με τους κατεξαίρεση εταίρους μας Ισλανδία και Νορβηγία. Άρα λοιπόν χαιρόμαστε πολύ για την συμμετοχή των δύο αυτών χωρών στο Σέγγεν. θα μπορούσαμε να πούμε εδώ ότι έκλεισε ο κύκλος. Το σημείο κίνησης των διαπραγματεύσεων αυτών ήταν η έγκριση του εντάλματος, του Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης, που υιοθετήθηκε υπό Βελγική Προεδρία επίσης. Τότε δεν προχωρήσαμε περισσότερο, δεν ήταν ε, δυνατόν γιατί το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης δεν θεωρήθηκε ως κομμάτι του Σέγγεν, αλλά γι' αυτό χρειάστηκε να ξεκινήσουν οι πραγματεύσεις με τις δύο αυτές χώρες για να δούμε πώς θα μπορούσαμε να εφαρμόζουμε ένα αντίστοιχο σύστημα και στην Ισλανδία και την Νορβηγία έτσι ώστε και δύο αυτές χώρες να βρίσκονται πιο κοντά στον ε, μηχανισμό που προβλέπεται από το Ευρωπαϊκό Άντελμα Σύλληψης. Πάλι λοιπόν τώρα, υπό Βελγικής Προεδρίας, έχουμε μπροστά μας τις συμφωνίες αυτές που ελπίζουμε ότι θα καταλήξουν επί Βελγικής Προεδρίας. Πρόεδρος. Ο Κλοντ Μωράης δεν θα μπορέσει να έρθει από ό,τι μου λένε, οπότε την επόμενη φορά θα πρέπει να μπει το θέμα του στην ημερήσια διάταξη και τώρα θα δώσω το λόγο στον κύριο Ταβάρες. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ και την Επιτροπή και το Συμβούλιο για τις παρουσιάσεις τους. Άρα εξετάζουμε μόνο την συμφωνία που έχει να κάνει με το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης. Θέλω να ευχαριστήσω την Επιτροπή που μας εξήγησε γιατί πήρε τόσο πολύ χρόνο ώστε να έχουμε την συμφωνία αυτή. Χωρίς να μπούμε σε λεπτομέρειες για τα αίτια ή τις επιπτώσεις του Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης, θα θέλαμε περισσότερες πληροφορίες για την εφαρμογή του όμως. γιατί έτσι θα μπορούμε να ξέρουμε τα υπέρ και τα κατά της επέκτασης του Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης στην Ορβηγία και την Ισλανδία. Για παράδειγμα, πόσες φορές έχει χρησιμοποιηθεί το Ευρωπαϊκό αυτό ένταλμα, πόσες ε, προσφυγές έχουν προκύψει εξαιτίας του. Τέτοια πράγματα θα ήταν καλό να έχουμε στατιστικά στοιχεία γιατί και από την άλλη μεριά θα μπορέσουμε έτσι να αξιολογήσουμε και πόσο πολύ θα χρησιμοποιηθεί από την Ορβηγία και την Ισλανδία. Πριν να έχουμε το Ευρωπαϊκό Άνταλμα Σύλληψης και σε αυτούς, δουλεύαμε στα πλαίσια των διμερών συμφωνιών έκδοσης. Θέλω να ξέρω λοιπόν πόσες φορές έχει χρησιμοποιηθεί αυτός ο μηχανισμός έκδοσης με την Νορβηγία και την Ισλανδία. Έτσι θα ξέρουμε πόσο χρήσιμη είναι και η τωρινή επέκταση. Έχω μια συγκεκριμένη ερώτηση για κάτι στο οποίο αναφέρθηκε η Επιτροπή και αυτό είναι η εξαίρεση για την επανήλυση διπλής εγκληματικότητας, είτε από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε από πλευράς Νορβηγίας και Ισλανδίας. Αυτή η μερική εξαίρεση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εγκλήματα στο οποίο επιβάλλεται ποινή τριετής ή μεγαλύτερη. Και υπάρχει ένας κατάλογος που περιλαμβάνει τα παραπτώματα αυτά τα οποία υπόκειται σε αυτή τη ρύθμιση. Για παράδειγμα, μία περίπτωση στο άρθρο 3, αριθμός 4, Παύλα 13 που μιλάει για διευκόλυνση μίας εισόδου σε χώρα χωρίς να υπάρχει άδεια. Τι ακριβώς εννοείται εδώ. Εννοείται περιπτώσεις εμπορίας ανθρώπων, Ορισμένοι εδώ και εγώ είμαστε πολύ ευαισθητοποιημένοι στο θέμα της εμπορίας ανθρώπων. Άλλο αυτό όμως και άλλο η διευκόλυνση εισόδου. Τι ακριβώς εννοείται εδώ. Υπάρχει ήδη κάποια δήλωση για εξαίρεση επαλήθευσης διπλής εγκληματικότητας για αυτό το συγκεκριμένο θέμα, για αυτή τη συγκεκριμένη περίπτωση. Εάν όχι, η καθυστέρηση επιτρέπει στην ε, Νορβηγία και στην Ισλανδία να υποβάλει τώρα μια τέτοια δήλωση και αν υπάρχει ήδη μια τέτοια δήλωση, για ποια εγκλήματα. και για αυτό το συγκεκριμένο έγκλημα, διευκόλυνση δηλαδή μη επιτρεπόμενη εισόδου. Τι είναι αυτό, πρόκειται για λαθρεμπόριο ή όχι. Στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης έχει ήδη χρησιμοποιηθεί μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πού. Ξέρουμε κάτι. Αυτή είναι λοιπόν μια συγκεκριμένη ερώτηση που έχω. Κατά τα άλλα, ευχαριστώ πολύ την Επιτροπή και το Συμβούλιο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Αυτή ήταν πολύ καλή ενημέρωση και θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Γκράντα εάν θέλετε να απαντήσετε σε αυτό το θέμα. Thank you, Madam Chair, and thank Της διπλής εγκληματικότητας. Του διπλού δεδικασμένου. Ναι. Θα προσπαθήσω να απαντήσω. Τα, στα δύο τελευταία ημερολογιακά έτη, εξαιρώ το παρόν, το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης ε, χρησιμοποιήθηκε για τα έτη 2008 και 2009 14.000 φορές. Κάθε χρόνο, κάθε έτος από τα δύο αυτά φαίνεται, διαφαίνεται ότι φέτος θα ξεπεράσουμε αυτό τον αριθμό. Όταν ερχόμαστε στο θέμα των σχέσεων με την Ορβηγία και την Ισλανδία, αυτό που μας ζητάτε κύριε Ταβάρες να κάνουμε είναι μία πρόγνωση για το μέλλον. Και δεν θέλω να υπησέλθω σε τέτοιες εικασίες αυτή τη στιγμή έχοντας υπόψη τα στοιχεία απελάσεων ε, από την Ισλανδία και την Νορβηγία έχουν υπάρξει προηγούμενα και έχουν υπάρξει περιπτώσεις. Η νομική βάση που έχει χρησιμοποιηθεί πολλές φορές είναι η σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης του 1955 όσον αφορά τις απελάσεις. Ε, το 1957, συγγνώμη, η Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για το 1957 για τις απελάσεις αυτό που πιστεύω ότι θα γίνει είναι ότι αυτές οι συμφωνίες θα χρησιμοποιηθούν όλο και περισσότερο δεδομένου ότι ζούμε σε μια εποχή μεγάλης κινητικότητας πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, του ΕΟΧ. Με αυτήν την αυξημένη λοιπόν κινητικότητα θα υπάρξει και μεγαλύτερη ανάγκη προσφυγής σε αυτήν την ταχύτερη διαδικασία παράδοσης ε, των κατηγορουμένων ε, μέσα στα πλαίσια της έκδοσης τους. Όσον αφορά αυτό του διπλού δεδικασμένου, δεν θα ήθελα να σταθώ σε αυτό το σημείο για να μην μακρηγορήσω. Όμως, σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε να διευκρινίσω πώς λειτουργεί το σύστημα αυτό του double criminality. Σας παραπέμπω στο άρθρο 6 να το μελετήσετε. Υπάρχουν δύο Is about a mandatory waiver of double criminality. Διατάξεις στο άρθρο 3. Η πρώτη Which we have... καλύπτει μία εξαίρεση του άρθρου αυτού με την συμφωνία, με την έναξη της συμφωνίας υπάρχει μία ρήτρα εξαίρεσης από το άρθρο αυτό της, ε, του double criminality. Απ' την άλλη πλευρά, όταν ε, δούμε το, την παράγραφο 4 του άρθρου 3, έχουμε μία προαιρετική εξαίρεση, εξαίρεση. Γιατί είναι προαιρετική, διότι συνδέεται με μία δήλωση η οποία θα πρέπει να γίνει από την Ορβηγία και την Ισλανδία ξεχωριστά δηλαδή και από την άλλη πλευρά από το συγκεκριμένο το ενδιαφερόμενο κράτος ε, μέλος μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάθε κράτος μέλος χρειάζεται να ζητήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνει μια δήλωση εκ μέρους του για την εφαρμογή αυτής της προαιρετικής ρήτρας. Τι γίνεται αυτή τη στιγμή. πρόσφατα εξέτασα αυτό τον κατάλογο και Κανένα κράτος, εκτός από την Αυστρία, δεν έχει κάνει ένα τέτοιο αίτημα να γίνει μια δήλωση εκ μέρους της χώρας μέσω Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η, Αυστρία, η Αυστρία έχει ζητήσει την έναρξη αυτής της διαδικασίας δήλωσης. Η Ισλανδία και η Νορβηγία δεν έχουν ξεκινήσει τη διαδικασία. Αναμένουμε από την Νορβηγία να ξεκινήσει τη διαδικασία, δεν ξέρουμε αν η Ισλανδία το κάνει δεν υπάρχει προθεσμία. Αυτέ, ε, αυτές οι δύο συμφωνίες ε, δεν προϋποθέτουν ε, προθεσμία. Όποτε θεωρήσουν την εποχή κατάλληλη, μπορούν οι χώρες αυτές να ξεκινήσουν τη διαδικασία δήλωσης, δημοσίευσης της δήλωσης και πιστεύω ότι καλό θα είναι να αποφασίσουν το ταχύτερο, γιατί οι πορείες θα ακολουθήσουν. Και τελευταία θα απαντήσω την πιο δύσκολη ερώτηση. Τι εννοούμε με αυτήν την διευκόλυνση ε, παράνομης ε, εισόδου και παραμονής. Καταρχάς, κάθε μέσον το οποίο βασίζεται στην αμοιβαία αναγνώριση καλύπτει τέσσερις βασικές ε, ε παραβιάσεις ε, οι οποίες καλύπτονται με την αμοιβαία αναγνώριση των ε, ποινικών πράξεων. Τι γίνεται τώρα με το θέμα της ε, ε, παράνομης διακίνησης ε, ανθρώπων σε σχέση με την παράνομη είσοδο. Ενδεχομένως η... domestic law. No need for... Ναι, η εμπορία ανθρώπων μπορεί να διέκοψε ο ε, ε, έκλεισε το μικρόφωνο του μιλητή. Ε, ενδεχομένως η εμπορία ανθρώπων μπορεί να συνδυαστεί με, την παράνομη, με το θέμα της παράνομης εισόδου και διαμονής. Όμως, στο θέμα της εμπορίας ανθρώπων, πρέπει να εξετάσουμε το ευρύτερο πλαίσιο και το μικρότερο πλαίσιο. Προηγούμενα δεν υπάρχουν στο εσωτερικό επίπεδο το, ευρωπαϊκό το, το, το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων δεν είχε μέχρι τώρα την ευκαιρία να εκδώσει απόφαση για αυτή τις συγκεκριμένε ε, ποινικέ πράξεις. Δεν υπάρχει λοιπόν προηγούμενο στην εσωτερική επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ, λέει Πρόεδρος, πριν ολοκληρώσουμε. Να ρωτήσω αν έχετε σχόλια. Oui, euh, merci. Euh. Ευχαριστώ πολύ που μου ξαναδίδετε το λόγο. Πιστεύω ότι η Κομισιό απήντησε στις ερωτήσεις που ακούστηκαν. Αυτό το οποίο θα μπορούσα να διευκρινίσω από πλευράς της Προεδρίας είναι ότι η συμφωνία του 2006 προσφέρει κάποιες δυνατότητες ε, δήλωσης. Υπάρχουν όμως και κάποιες χώρες που ακόμα δεν έχουν ε, δηλώσει στο Συμβούλιο τις ε, προθέσεις του σχετικά με αυτές τις δυνατότητες δηλώσεων. Έχουμε στείλει μια, μια υπενθύμηση και ελπίζουμε ότι άμεσα θα έχουμε στη διάθεσή μας τις δηλώσεις των κρατών μελών και μετά θα μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε τη σύναψη της συμφωνίας. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ για αυτή την τόσο ενδιαφέρουσα συζήτηση. Δεν... Α, θα θέλετε να προσθέσετε κάτι, θέλετε να απαντήσετε κάτι, ο κύριος Ταβάρες. Να ρωτήσω το Συμβούλιο προβλέπονται κάποια χρόνια για τις ε, διμερείς συμφωνίες έκδοσης ε, Ισλανδίας, Νορβηγίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης από την άλλη. Ε, για να έχουμε μια εικόνα της πραγματικότητας. Okay, thank you very much. Since we don't have any other... Ωραία. Λοιπόν, μια και δεν υπάρχει τίποτα άλλο στα διάφορα. Α, όχι, όχι, όχι. Α, ναι, να απαντήσουμε. Ναι, ναι, ναι, ναι. Όντως, πρέπει να δοθεί μια απάντηση. Ναι, ναι, ναι. Ζητώ, συγγνώμη πρόεδρε. Δεν θέλω απάντηση τώρα, γραπτά, να μου πείτε αν, πότε έχει χρησιμοποιηθεί η συμφωνία αυτή. Ε, ούτως ή άλλως, μια και δεν ξέρουμε και τις αντιδράσεις των κρατών μελών, θα επανέλθουμε στο θέμα αυτό. Μην ανησυχείτε. Λοιπόν, η συμφωνία της επο... η... η επόμενη συνεδρίασή μας ε, θα είναι στις 15 Νοεμβρίου το απόγευμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ ε, όλους για τη συνεργασία σας.